σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων ε, μέτρων κατά τη φοροαποφυγή και του ξεπλήματο χρήματο ε, υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων ε, για το Panama Papers. Το λόγο λοιπόν έχει η κυρία Υπουργό Ένι Πλάσχαρτ. Ευχαριστώ εκ νέου κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Όσον αφορά τα Panama Papers, να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλα αυτά αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά την ανάγκη να συνεχίσουμε την καταπολέμηση των φορολογικών απατών και του ξεπλήματος χρήματος. Είναι πολύ πρόημο τώρα να προβούμε σε πλήρη ανάλυση του σκανδάλου Panama Papers, αλλά όλοι μας εξετάζουμε τις συνέπειες και τις απαντήσεις που πρέπει να βρεθούν. Οι εθνικές κυβερνήσεις ανακοίνωσαν έρευνες συζητώντας το που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνω μια διάκριση μεταξύ του κειμένου ε, και μάλλον του φορολογικού κομματιού και του ξεπλήματος χρήματος από την άλλη. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε δύο πορείες. Χρειαζόμαστε πρώτα σε πληροφορίες και δεύτερον χρειαζόμαστε μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για να καταπολεμηθούν οι απάτες. Το πακέτο καταπολεμήσεως φοροαπηφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο. Σημαντική βάση για να εφαρμοστούν διεθνείς προδιαγραφές και να συμπεριληφθούν στη δική μα νομοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση πληροφορίε, υπάρχουν διεθνεί προδιαγραφέ για τη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών και έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΣΑ. Σημαντική πρόοδο έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, όμω όχι όλοι οι διεθνεί παίκτε έχουν δεσμευτεί ακόμα να παίξουν ένα δίκαιο παιχνίδι και αυτό ισχύει κυρίω για τον Παναμά. Για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική διαφάνεια για τα φορολογικά, πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μεγάλος παίκτη διεθνής πρέπει να μιλά με μια φωνή και να πείσει τους εταίρους της στο διεθνές προσκήνιο να εθετήσουν τα συμπεφωνημένα πρότυπα που τα στήριξε η πλειοψηφία. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουν προχωρήσει και πιο πέρα από τα πρότυπα όσα και πολλοί μας θεωρούν σαν επικεφαλής και αυτό είναι καλό. Υιοθετήσαμε μια οδηγία για διοικητική συνεργασία που συμπληρώθηκε πρόσφατα ούτως ώστε να καλύπτει και την ανταλλαγή αποφάσεων tax rulings και μετά θα έχουμε κατά χώρα εκθέσεις που θα υποβάλλεται από τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πακέτο πρότεινε. Στο Συμβούλιο έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά τις εκθέσεις κατά χώρα και, και παροτρύνω μάλλον και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εθετεί στην γνωμοδότησή του ταχύτερο δυνατόν. Βεβαίω δεν θα σταματήσουμε εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σήμερα μια πρόταση για δημόσια έκθεση κατά χώρα όσον αφορά τι πολυεθνικέ, ε, αύξηση τη διαφανεία και αυτή η πρόταση θα τύχει τη πλήρου προσοχή του Συμβουλίου. Όσο αναμένεται η Προεδρία, σίγουρα θα προσπαθήσει ούτω ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση. Επανερχόμενοι τώρα σε αποκαλύψει. Θέλω να αναφερθώ στο τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από την αύξηση ανταλλαγή πληροφοριών, ούτω ώστε να καταπολεμήσουμε τη φορολογική απάτη και τη φοροαποφυγή, καθώ και το ξέπλυμα χρήματο. Τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση για εξωτερική στρατηγική για αποτελεσματική φορολόγηση σαν τμήμα του πακέτου για την καταπολέμηση φοροαποφυγή. Προτείνουμε κοινό κατάλογο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, σχετική διαδικασία για να, απαντάμε σε, να ανταποκριθούμε σε τέτοιε χώρε που δεν σέβονται με τα πρότυπα για τη σωστή φορολόγηση. Η Προεδρία προσπαθεί να αντιδράσει γρήγορα στον αφορά τι προτάσει και να λάβει υπόψη και την περίπτωση των Panama Papers. Τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πακέτο της περιείχε και πρόταση οδηγίας που καθορίζει κανόνες κατά της φοροαποφυγή και των πρακτικών. Την οδηγία για την φοροαποφυγή η οποία εξετάζεται τώρα που μιλάμε. Κάποιοι από τους κανόνες του σχεδίου οδηγίας θα μπορούσαν να είναι κρίσιμοι διότι μιλάμε και για καταχρηστικές μορφές φοροαποφυγή. Χρειάζεται νόμιμη φοροαποφυγή. Άρα Πρέπει να προωθηθεί το μέτρο ταχύτερο δυνατόν. Προσπαθούμε να πετύχουμε συμφωνία από τη προτάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βασιστούμε στην υποστήριξή σα, στη στήριξη του Κοινοβουλίου. Τέλο, να σε επιστήσω την προσοχή στο έργο που γίνεται από την ομάδα του Κώδικα Διντολογία Επιχειρήσει και να αποφευθούν ε, τα επιβλαβή καθεστώτα φορολόγηση. Θέλει ο, οι αρχέ να υιοθετηθούν σε τρίτε χώρε. Εργάστηκε επιτυχώ στην Ελβετία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητούμε με το Λίχτενστάιν εκ μέρους της ομάδας και συνομιλούμε και με άλλες χώρες. Μάλλον θα πρέπει να συμμετάσχουν και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, να στραφώ εντάχει στο ξέπλυμα χρήματος. Αυτό το θέμα συνδέεται στενά με τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας και έχει ύψιστη προτεραιότητα για μας το Φεβρουάριο, σε αντίδραση του σχεδίου δράση για την καταπολέμηση τη χρηματοδότηση των τρομοκρατών, το Συμβούλιο συμφώνησε να προχωρήσει γρήγορα με την εφαρμογή σειρά μέτρων τα οποία θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση και τη χρηματοδότηση των τρομοκρατών και του ξεπλήματο του χρήματο. Να περιγράψω τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τη συζήτησή μα τη σημερινή. Πρώτα απ' όλα οι Υπουργοί τόνισαν την ανάγκη για εντοπισμό των τρίτων χωρών εκείνων που έχουν στατηγικά ελλείμματα όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματο ε, και τη χρηματοδότηση των τρομοκρατών. Έχουν κενά. Θα γνωρίζετε σύμφωνα με το με την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα συμμόρφωση όσον αφορά τι χρηματοπιστωτικέ ροέ από και προ τι χώρε που είναι στον κατάλογο. Το Φεβρουάριο ζητήσαμε να ολοκληρωθεί ο εντοπισμό μέχρι, το τέλος, μέχρι αρχέ Μαΐου. Εδώ είμαστε στα χέρια όμω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, βιάζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εργάζεται σκληρά για το θέμα. Ελπίζουμε ότι τελικά να συμφωνεί και το Κοινοβούλιο και να κινηθεί ταχιστά. Δεύτερον, οι Υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία που έχει η επιτάχυνση. Η εφαρμογή του πακέτου πολέμηση του ξεπλήματος του χρήματος. Κάτι που το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο θέτησαν πέρσι. Κοινό στόχος. Ολοκλήρωση της διαδικασία. Και αυτό μέχρι τέλος του έτους. Τρίτον, αναλάβαμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και των διάφορων ε, υπηρεσιών των υπευθύνων οικονομικά και ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέχρι τον Ιούνιο κάποιου στόχου, κάποιε βελτιώσει όσον αφορά την οδηγία την τέταρτη για το ξέπλυμα χρήματο. Ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να εισαχθούν και όρια σε μεγάλε πληρωμέ σε ρευστό και μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξεταστούν ενδεχόμενα μέτρα για χαρτονομίσματα ε, υψηλή αξία όπω το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Η οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματο ε, χρήματο είναι πολύ πρόσφατη και ακόμα είναι καθοδόν όσον αφορά τη συμπερίληψη ενόμη τάξη των κρατών μελών. Όμω, ήδη έχει καταστεί σαφέ ότι στοχευμένε τροπολογίε χρειάζονται να ενισχύσουμε την πρόσβαση στις πληροφορίες Φερρυπίν. Πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικής και πληρωμών από τις μονάδες υπεύθυνες για τα οικονομικά, δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Να εντοπιστούν οι τρίτες χώρες που είναι επικίνδυνες ε, και τι γίνεται και με τα εικονικά νομίσματα. Το Συμβούλιο θα επεξεργαστεί προς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι θέμα προτεραιότητας και σίγουρα αυτό θα είναι κάτι που θα ισχύσει και για το Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρω ότι το θέμα του ξεπλήματο χρήματο και τη χρηματοδοτή των τρομοκρατών έχει στην προτεραιότητα και στη διεθνή μα ατζέντα, κυρίω στα πλαίσια τη ομάδα κρούση για τα χρηματοστικά θέματα και στου G20. Κλείνοντα, Πρόεδρε, να πω ότι η Προεδρία αποφάσισε τα Panama Papers να τα βάλει στην ημερήσια διάταξη του ατύπου Εκοφίν στο Άμστερνταμ στις 22 Απριλίου, εκεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να αντιδράσει όσον αφορά την επισκόπηση των πρωτοβουλειών για την καταπολέμηση ξεπλήματος χρήματος και τη φορολογική απάτη. Οι υπουργοί και οι διοικητές κεντρικών τραπεζών θα ανταλλάξουν απόψεις. Και προσβλέπω σε αυτή τη συγκεκριμένη ανταλλαγή των απόψεων και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ και τώρα το λόγο έχει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο, ο Επιτρόπος Μοσκοβισή. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά που δίνει μια νέα και βελτιωμένη ε, νομοποίηση στο πρόγραμμά μας ε, κατά τη φοροδιαφυγή και τη νομοποίηση εισόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Αν κανεί ήθελα αποδείξει για το πόσο σημαντική είναι η κοινή μα δουλειά στον τομέα αυτό, τι έχει και είναι γνωστέ στη σπάση. Με το εξωσημείο το έργο που θέλω να το επισημάνω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μόνο με τη διαφάνεια και την καλή φορολογική και δημοσιονομική διακυβέρνηση και είναι μέτρα που τα ζητούμε εδώ και καιρό. Ε, αν αυτά είχαν εφαρμοστεί ε, και σε διεθνή κλίμακα, αυτή η ε, αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, ε, αυτή η συγκάλυψη, ε, αυτή οι κρυφοί λογαριασμοί δεν θα ε, υπήρχαν. Πραγματικά ήταν τεράστιες συγκλονιστικές αυτές οι αποκαλύψεις αλλά και πάρα πολύ επιζήμιες. Οι πολίτες μας δεν μπορούν να κατανοήσουν ούτε να αποδεχθούν τις πρακτικές αυτές που τελικά στην πράξη συνιστούν κλοπή. Ας, μην τολμήσουμε, να την πούμε αυτή τη λέξη. Αυτό που ε, βιώνουμε είναι αυτή η δημόσια γανάκτηση και πρέπει ε, να την, μετατρέψουμε σε ευκαιρία και να δράσουμε. Αυτή είναι η ευκαιρία που μας προσφέρουν αυτές οι αποκαλύψεις, γιατί έχουμε πλέον μια ευκαιρία ως πολιτική, αλλά έχουμε και το καθήκον ε, ως πολιτική να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τη φοροδιαφυγή. Τη φοροαποφυγή και τη φοροαπάτη τις πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος. Είναι η ευκαιρία μας ε, να ενισχύσουμε ε, τη δυναμική του ήδη φιλόδοξο προγράμματό μα για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή τη νομοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε, ιδίω ζητώντα από τα κράτη-μέλη την πολιτική του δέσμευση να αντιμεταφράσουν σε δράση, σε συγκεκριμένα έργα και το ζητώ και από αυτό το βήμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτός ο μηχανισμός και θα πρέπει και να δούμε και τι νέα μέτρα μπορούμε να λάβουμε για να ενισχύσουμε την άμυνα της Ένωσης κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Επίσης είναι ευκαιρία για να εντείνουμε τη συνεργασία μας με τους διεθνείς εταίρους για να ασκήσουμε πιέσεις σε προβληματικές δικαιοδοσίες, φορολογικούς παραδείσους όπως τους αποκαλούμε για πιο ε, δίκαιη διαφανή ε, φορολογία σε διεθνές επίπεδο. Και θα ζητήσουμε από τις χώρες αυτές να ακολουθήσουν τα δικά μας πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Ε, μια λέξη για όσα έχουν γίνει, γιατί δεν θα πρέπει μόνο να κατηγορούμε αυτούς, έχουν γίνει και πολλά θετικά. Παραδείγματος χάρη, μεγαλύτερη διαφάνεια Προσπαθούμε να ανακτήσουμε βέβαια το χαμένο έδαφος, αλλά δεν ξεκινάμε και από το μηδέν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πολύ στεναρές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος και για τις επιχείρησεις και για τους απλούς πολίτες και πράγματι τους τελευταίους μήνες καταθέσαμε ούτε λίγο ούτε πολύ τρεις δέσμες ε, μέτρων. Ε, πρώτον, μία πρόταση που περιλάμβανε νομικώς δεσμευτικά μέτρα κατά της φοροαποφυγής. Προβλέπει και το γενικό κανόνα κατά των καταχρήσεων, ώστε δομές offshore, εξωχώριες τεχνητές δομές, να ε, χρησιμοποιούνται για φοροαποφυγή. Και από την άλλη επιβάλλονται κανόνες στις εταιρείες της Αλοδαπής, Control Foreign ε, Corporate Rules λέμε ε, στα αγγλικά, ώστε αυτή, αυτά τα φορολογικά έσοδα να μην χάνονται. Γιατί πολλές φορές δεν φορολογήθηκαν τα έσοδα πολλών ε, εταιριών ή ε, φορολογήθηκαν με μια πάρα πολύ ευνοϊκή φορολογική βάση. Και τα βλέπουμε και στα έγγραφα του Παναμά. Δεύτερον, έχουμε καταθέσει φιλόδοξες προτάσεις ε, για περισσότερη φορολογική διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών μεταξύ κρατών μεταξύ επιχειρήσεων ε, και φορολογικών διοικήσεων. Και τρίτον, επίσης, βελτιώνουμε τη φορολογική διαφάνεια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτε ευρωπαϊκές χώρες καταρχά και χαίρομαι πολύ που καταφέραμε να υπογράψουμε, τέλο πάντων διαπραγματευτούμε, να συνάψουμε συμφωνίε με την Ελβετία, το Λίχτεστάιν, το Σαν Μαρίνο, Ανδόρ, ε, Μονακό, ε, σύντομα, Δημερεί συμφωνίε με πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τους πολίτες μας. Το τραπεζικό απόρριτο πνέει τα λίστια πλέον στην Ευρώπη και αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Αλλά και εκτός Ευρώπης ε, είχαμε τις προτάσεις για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού κοινού καταλόγου φορολογικών παραδείσων στο πλαίσιο της εξωτερικής μας στρατηγικής για αποτελεσματική φορολόγηση, την κατέθεσα τη σχετική πρόταση τον Γενάρη. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων κατά της ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής και το συζητά αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο αυτό το πακέτο. Αυτές λοιπόν είναι οι νέες πρωτοβουλίες ε, γιατί ζητήθηκε διαφάνεια και αυτό ισχύει ήδη για ε, τους, ε, ε, τους τραπεζικούς λογαριασμούς στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και από το 2017 θα έχουμε αυτόματη ανταλλαγή πολλών πληροφοριών των τραπεζών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ώστε να μην μπορούν οι φοροδιαφεύγοντες να κρύβουν τις οικονομίες και τις απειταμιεύσεις τους σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Πριν από λίγα λεπτά αποφάσισε η Κομισιόν ε, το όριο αυτής της φορολογικής διαφάνειας να το βάλει ακόμη πιο μακριά. Δηλαδή οι διεθνείς όμιλοι πλέον θα πρέπει ε, να δημοσιοποιούν ε, το reporting των δραστηριοτήτων τους αναχώρα. και θέλω να σας τα πω όλα αυτά γιατί θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από την αρχή πραγματικά ήμουν υπέρ αυτής της δημοσιότητας, της δημοσιοποίησης όλων αυτών των στοιχείων και χαίρομαι πολύ που σήμερα η Κομισιόν προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το λέω σε όσους θα υποστηρίξουν ότι δεν είναι αρκετά όλα αυτά, να γίνει η πρώτη οικονομική ζώνη στον κόσμο που δημοσιοποιεί αναχώρα τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, των ομίλων. Ε, κουνάτε το κεφάλι σας κύριε Λάμπερτς, αλλά ξέρετε όπως και εγώ ότι ο ΩΣΑ πρότεινε να υπάρξει ένα όριο, ε, και αυτό δεν αμεληταίο, ε, στις ανταλλαγές μεταξύ φορολογικών προς το παρόν. Έτσι. Ξέρω ότι κάποιοι ε, διαρωτάστε σε αυτό το όριο που ουσιαστικά ε, θα μας βοηθήσει να λέμε το 80% των δραστηριοτήτων. Λέτε όμως και γιατί εκτός της Ευρώπης δεν υπάρχει κάτι. Θέλω να σας πω ότι πρώτον με ομαδοποιημένα στοιχεία θα προχωρήσουν και για τις άλλες περιοχές του κόσμου και κάτι ακόμη. Ε, θα δώσουμε και αναλυτικά στοιχεία για τις δραστηριότητες διεθνών ομίλων που έχουν δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους δεν μπορούν να ξεφύγουν. Είναι σημαντικά όλα αυτά και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικροτήσει τι προσπάθειε, αλλά σίγουρα θα συνεχίσουμε από κοινού τι προσπάθειε μα. Έχουμε λοιπόν σημαντική πρόοδο σε κάποια μέτωπα με τι φορολογικέ μα πρωτοβουλίε, η γρήγορη συμφωνία για δύο προτάσει περί διαφάνεια. Βέβαια, πολλά σημαντικά μέτρα είναι ακόμη επιτάπητο στο Συμβούλιο. Τα έγγραφα του Παναμά είναι ένα μήνυμα προ τα κράτη-μέλη να δείξει το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας με την Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο, ε, καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή, συμφωνώντας σε νέες διατάξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα μας κατά του ξεπλήματος χρήματος. Τα κράτη-μέλη οφείλουν οφείλουν πάση θυσία να ε, αναλάβουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις, ε, να τις υλοποιήσουν. Ε, συγκεκριμένα έχουμε την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που πρόλειπε μεταξύ άλλων την ταυτοποίηση των πραγματικών ιδιοκτητών εταιρεών και τράστα και τη δημιουργία εθνικών μητρών. Πρέπει να εγκριθεί και να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο αυτή οδηγία. Το ζητούμε εδώ και καιρό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μα θα βοηθήσει να αποτρέψουμε την κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματο για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Η Κομισιόν θα δώσει τη δέουσα υποστήριξη για να διευκολύνει τη διαδικασία μεταφορά αυτή τη οδηγιά σε εθνικό, στο εθνικό δίκαιο και για την ορθή μεταφορά των διατάξεων αυτής της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ, και στρέφομαι και προς την ε, Προεδρία του Συμβουλίου ότι πρωταρχική ευθύνη να πω και στα κρατημέλη. Αυτό το μήνυμα των Panama Papers, αυτό το μήνυμα που στέλνετε κι εσείς ε, ως Κοινοβούλιο και το μήνυμα της Κομισιόν ε, πρέπει να εισακουστεί και πρέπει τα κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι δεν μπορούν στον τομέα αυτό να επιδεικνύουν υπερβολική σύνεση και εποπτεία. Όλοι πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις. Τι άλλο πρέπει να γίνει ακόμη όπως είπα ήδη έχουν γίνει πολλά. Έχουμε επιτυχίε στη μάχη κατά τη φοροδιαφυγή και του ξεβλήματο χρήματο. Όμω οι πρόσφατε αποκαλύψει δείχνουν ότι ακόμη απομένουν να γίνουν πολλά αν θέλουμε να περιορίσουμε τι τρευλώσει των διαφορετικών νομοθεσιών και αν θέλουμε να συνεργαζόμαστε απόλυτα και πλήρω μεταξύ μα. Ένα τομέα κλειδί ε, στον οποίο χρειάζεται περισσότερη δουλειά είναι αυτό. Και βέβαια Υπάρχουν ακόμη πολλές διατάξεις και προτάσεις που συζητούνται σε επίπεδο Συμβουλίου αυτή τη στιγμή και που θα περάσουν τα μάλα. Ε, παραδείγματι, η οδηγία κατά της φόρο διαφυγής. Επιθυμώ, το γνωρίζω και εγώ όπως και η Ολλανδική Προεδρία, ότι ε, πρέπει να θέλουμε να εγκριθεί. Πριν το καλοκαίρι είπατε κυρία μου ότι το ΕΚΟΦΗΝ, το άτυπο ΕΚΟΦΗΝ, ε, συνεργάζεται στις 22 ε, Απριλίου και θέλουμε να τεθεί επιτάπητος όλο το πακέτο συνολικά και εποφελούμε για να πω σε κάποιους υπουργού που λένε ότι θέλουμε το μισό. Αν έχουν το μισό ε, πακέτο θα έχουν και τα μισά αποτελέσματα. Όχι, δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε ημίμετρα. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι τέλους. Πρέπει να καταπολεμήσουμε, ε, πρέπει να φτιάξουμε ένα κατάλογο, ένα μαύρο κατάλογο, ε, μια μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων. Ήδη η Κομισιόν έχει ένα κατάλογο, έχει μια λίστα που είναι ένα είδος συμπιλήματος ε, των καταλόγων των εθνικών που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Η Πορτογαλία έχει 85 φορολογικούς παραδείσους στη λίστα. Μήπως είναι πολύ. Η Γερμανία δεν έχει κανένα. Είναι πολύ λίγο αυτό. Και άμα πάρω το παράδειγμα του Παναμά, σε παγκόσμιο επίπεδο ε, είδαμε πόσο είναι φορολογικό παράδεισο η χώρα αυτή και ελπίζουμε να αλλάξει εκεί η κατάσταση. Οκτώ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εννέα από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί προσθέθηκε η Γαλλία, που έτσι. Πολύ λίγε χώρε λοιπόν, άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα πανευρωπαϊκό κατάλογο φορολογικών παραδείσων. Έξι μήνε βάζω εγώ ω διορία για τις καλές μεθόδους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ε, σύντομο το αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και επίσης πρέπει να ενισχύσουμε και το κανονιστικό πλωστάσιό μας. Για παράδειγμα, ήδη ανακοινώσαμε την αναθεώρηση της οδηγίας κατά της νομιμοποίησης όλων από δραστηριότητας για τον Ιούνιο. Και θα πρέπει σίγουρα να διδαχθούμε και από τις αποκαλύψεις ε, των εγγράφων του Παναμά υπάρχει και μια πολύ σημαντική διάσταση, η διεθνή διάσταση. Διότι φυσικά είναι από τη μία αυτά που έχουμε να κάνουμε εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι ήδη προηγείται σε σχέση με άλλε χώρε, με άλλε περιοχέ του κόσμου. Είναι ε, ατμομηχανή και ηγέτη ε, στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, ό,τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι και πιο αποτελεσματικό φυσικά. Και γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο τη ομάδα των 20, του G20, πρέπει να προτείνουμε ένα νέο στάδιο, μια νέα φάση. Από την Πέμπτη, οι Υπουργοί Οικονομικών ε, του πλανήτη θα είναι στην Ουάσιγκτον για την Αρινή Σύνοδο του Νουτού. Και εκεί θα γίνει και μια συνεδρίαση του G20 σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών. Θα είναι εκεί και η Κομισιόν και θα προτείνουμε να πάμε πιο πέρα. Βλέπω πολύ ικανοποίηση, διότι ορισμένοι υπουργοί ε, χωρών μελών ε, του G20 θέλουν να μας ακολουθήσουν. Θέλουμε να μιλάμε με μία φωνή. Ήθελα με την εισαγωγή μου αυτή, αγαπητοί βουλευτές, να σας αναφέρω ποια είναι τα πρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαμε να θετήσουμε για να βελτιώσουμε την, ε, σε αυτές τις αδιαφανείς δομές, ανώνυμες συναλλαγές και όλα αυτά που ε, βγήκαν ε, στο φως με τις πρόσφατε αποκαλύψεις η Κομισιόν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να βασιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα δώσει ε, τροφή στη συζήτηση, θα μας πιέσει να ακολουθήσουμε τα επόμενα ε, στάδια σε αυτή τη διαδικασία και ελπίζω ε, ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι μπορείτε να βασιστείτε στην Κομισιόν. Είμαστε φυσικοί σύμμαχοι, μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις, αποχρώσεις, αλλά νομίζω ότι έχουμε τους ίδιους στόχους και αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε χέρι-χέρι με τις ευαισθησίες ε, μας ο καθένας, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Τόσο μακριά όσο μας ζητά ο Ευρωπαίος πολίτης, ώστε να έχουμε διαφάνεια και να μπορέσουμε αυτές τις πρακτικές ε, που σκανδάλισαν τον πλανήτη να ε, απαλληφούν. Και σήμερα και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Αν είχα την εντύπωση ότι μου λείπε δουλειά, για τα φορολογικά μέχρι το τέλος εντολής μου. Όχι μόνο πλέον ε, έχω δουλειά πολύ μπροστά μου ε, που δεν ξέρω αν θα μου φτάσει και τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πιτροπέ. Και τώρα το λόγο έχει ε, από πλευράς του ΕΛΚΟ ο κύριος Άλμπα Μπυρικαΐν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Οι πολίτες αρχίζουν πλέον να κουράζονται. Ευθύνη μας είναι να αποφύγουμε ε, να μας βλέπουν ως πρόβλημα. Και αντίθετα πρέπει να τους κάνουμε να μας βλέπουν ως λύση. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί στη δράση μας. Οι αποκαλύψεις ε, των εγγράφων ε, του Παναμά μας δείχνουν ακόμη μια φορά την ανάγκη να συνεχίσουμε να προχωρούμε όπως κάναμε και κατά το τελευταίο έτος με στόχο τη μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια. Το είπε και ο Επίτροπος. Έχουμε μια ευκαιρία, πολιτική ευκαιρία μπροστά μας και δεν πρέπει να την απολέσουμε. Μην έχετε αμφιβολία κύριε Επιτροπέ, θα σας στηρίξουμε. Θα σας στηρίξουμε σε όλα τα μέτρα τα οποία προτείνετε σήμερα εδώ ενώπιόν μας και θα στηρίξουμε και όλα τα μέτρα που θα προτείνετε στο μέλλον για να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα την φοροδιαφυγή. Διότι πραγματικά είναι αναγκαίο να ε, συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να τα αντιμετωπίσουμε. Και όπως είπατε δεν είναι αποκλειστικό ε, πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μια απάτη σε παγκόσμιο επίπεδο και με όσο το δυνατόν ε, περισσότερες χώρες συμμάχους σε αυτόν τον αγώνα. Φυσικά το να δημιουργηθεί μια εταιρεία από κάποιον στον Παναμά δεν είναι παράνομο. Παράνομο είναι τι κάνει κάποιο με αυτή την εταιρεία εκεί. Και αυτή είναι δική μα ευθύνη. Δηλαδή να αποφύγουμε τέτοιε εταιρείε ε, να τις χρησιμοποιούν κάποιοι για να φοροδιαφύγουν. Το ΕΛΚΑ πάντοτε προάσπιζε, θα προασπίζει δε και πάντοτε τη μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια. Το ΕΛΚΑ ζητεί. Η και οι κυβέρνηση του Παναμά να έρθουν ε, να καταθέσουν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχουν κάνει οι επιχειρήσει, το έχουν κάνει και άλλα κράτη στην Επιτροπή Τάξε. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση του Παναμά θα θελήσει να συνεργαστεί μαζί μας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τόσα δικηγορικά γραφεία ή κράτη να χρησιμοποιούν ε, ως διαπραγματευτικό μοντέλο αυτό τον φορολογικό σχεδιασμό για να ζουν σε βάρος άλλων κρατών. Πάρα πολύ καλά ε, ορίσατε τα πράγματα κύριε Επίτροπε. Πρόκειται πραγματικά περικλοπής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Σάλπα και τώρα ο Πρόεδρος Πιτέλα για το λόγο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε δισεκατομμύρια ευρώ που αφαιρούνται από το δημόσιο κουρβανά. Πολύ συχνά κυκλωμένο χρήμα που είναι ε, προϊόν παρανόμων δραστηριοτήτων εντός του των οποίων κρύβεται η μαφία, περί αυτού πρόκειται. Και αυτή είναι η χειρότερη όψη του χρηματοπιστωτικού μας καπιταλισμού, του διεφθαρμένου και του μολυσμένου από τους απαταιώνες. Γι' αυτό σας το λένε ονόματι των σοσιαλιστών και δημοκρατών, ανοχή μηδέν κατά εκείνων που φοραποφεύγουν, κατά των φορολογικών παραδείσων. Και γι' αυτό το λόγο εμείς θέλουμε να δημιουργηθεί μια επιτροπή έρευνας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, ούτως ώστε όλες ή δυνάμεις να διατεθούν για να σταματήσουμε τη διαφυγή. Να μην υπάρχει καμία δηλία όσον αφορά το σκοπό αυτό και μετριοπάθεια. Θέλουμε και μια διεθνή διάσκεψη, ε, μια παγκόσμια συνένεση που θα μπορέσει να ασχοληθεί με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Και μετά έχουμε και τα νομοθετήματα που ζήτησε ο Επίτροπος ο κ. Μοσκοβισή. Αυτό το σημείο ήταν στο επίκεντρο της της ε, συμφωνίας της ε, κυβερνήσεως και γι' αυτό υπερψηφίσαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κυρίου Γιούνκερ και ο Επίτροπος ο κ. Μοσχοβησή κινούνται με αποφασιστικότητα και σθένος. Όμως πρέπει να αποχωρήσετε πάρα πέρα. Να έχετε περισσότερο θάρρος και στην καταχώρα υποβολή εκθέσεων. Θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι χώρες του κόσμου δεν μπορούμε να περιοριστούμε. Είναι μια θετική προσπάθεια που δεχόμαστε με θικανοποίησος. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε πιο πέρα, να έχουμε μεγαλύτερο θάρρος έναντι ενός καρκίνου τόσο επικινδύνου, ενός ε, καρκίνου τόσο αρνητικού. Ζητάμε να κάνει και άλλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρχει ένα καθεστώς για τους πληροφοριοδότες και μια έκθεση για το Trade Secrets. Είναι ένα πρώτο βήμα ε, στη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε και πολιτικές δεσμεύσεις σε αυτή τη ενία. Χρειάζεται μια εναρμόνιση της φορολογικής βάσεως, της φορολογήσεως των εταιριών. Χρειαζόμαστε έναν ε, μαύρο κατάλογο των φορολογικών ε, παραδείσων και κυρώσεις κατά των επιχειρήσεων φοροαποφεύγων. Λοιπόν, προτεραιότητα αυτή τη θητεία θα πρέπει να είναι η εκρίζωση των φορολογικών παραδείσων και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Κοινοβουλίου. Έχετε μια ερώτηση από τον κύριο Κάζα. Θέλετε, δεχόσαστε. Ορίστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Πιτέλα, τον σέβομαι, είναι ειλικρινής πολιτικός, έχει ένα κέραιο. Συμφωνώ μαζί του ότι χρειάζεται να δείξουμε μηδενική ανοχή στους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο. Θα ήθελα ο κύριος Πιτέλα να μας πει πώς μπορούμε να περάσουμε στη δράση από τα λόγια. Έχουμε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση που αναμειγνύεται, έναν υπουργό από ε, ευρωπαϊκή χώρα και έναν επικεφαλής Υπουργικού Γραφείου χώρας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, είναι μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Όμως δεν θα πρέπει να κοιτάμε τα κόμματα τώρα, αλλά ποιο είναι το σωστό και εκείνο που πραγματικά είναι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω διακρίσεις και δεν κάνω εκπτώσεις. Εγώ δεν μίλησα για τον Κάνιατε. Το θέμα δεν είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το θέμα για πολιτικούς σκοπούς, αλλά πρέπει να είναι παντού να επικρατεί σαφήνεια. Θα πρέπει η σαφήνεια και το ξεκαθάρισμα να γίνει παντού, παντού. Σας ευχαριστώ και τώρα για το ECR. Το λόγο έχει, το λόγο έχει ο κύριος Λούκα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, Έχουμε εδώ ένα μεγάλο σκάνδαλο, αντίθετο θέμα και τα έγγραφα του Παναμά αποκάλυψαν αυτό που ήταν γνωστό σε όλους ε, και το θέμα είναι γιατί δεν είχαμε δραστηριοποιηθεί νωρίτερα. Ε, ναι. Έχουμε μία τρύπα και μπας νερό. Θα πρέπει να ρωτηθούμε πώς προέκυψε αυτή η τρύπα και ποιος ε, την άφησε να υπάρξει. Και υπάρχουν λοιπόν ε, πάρα πολλές δυνατότητες ε, για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής σε τέτοια μεγάλη κλίμακα. Θα πρέπει να ρωτήσουμε γιατί οι οικονομικές υπηρεσίες, ε, η εφορία δεν είχαν αντιδράσει ή μήπως το ήξεραν εδώ και καιρό ότι υπήρχε τέτοιου επίπεδου φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή και κατά πόσον το είχαν διαβιβάσει αυτό στους Υπουργούς Οικονομικών και το θέμα είναι γιατί δεν αντέδρασαν οι Υπουργοί Οικονομικών στην προκειμένη περίπτωση. Άρα έχουμε μια μεγάλη πολιτική αποτυχία και το ήξεραν αυτό οι κυβερνήσεις εδώ και καιρό. Όλοι, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ήξεραν ότι τέτοιου είδους φοροδιαφυγή λαμβάνει χώρα και τίποτα δεν έγινε. Αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα για τους φιλελεύθερους η κυρία Γκουλάχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Με χαρά βλέπω ότι η Ολλανδική Προεδρία μας στέλνει την Υπουργό Άμυνας. Θα επιτεθούμε κατά της φοροδιαφυγής με στρατιωτικά μέσα. Ίσως αυτό είναι κάτι καλό. Χαιρετίζω την παρουσία σας εδώ. Λοιπόν, πολύ πιο σοβαρά. Θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα επί το οποίο για την ομάδα των φιλελευθέρων δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Πρέπει να δράσουμε σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται μια δράση ερευνητική και νομίζω ότι είμαστε υπέρ και άλλε ομάδε ε, στο ημικύκλιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε στο έργο που έκαναν οι δημοσιογράφοι και του οποίου ετοίμησε και ο επίτροπο, να καταλάβουμε καλύτερα τι συνέβη, να εξακριβώσουμε κατά πόσο πραγματικά έχουμε όλε τι πληροφορίες. Είναι μια δουλειά ερευνητική πρέπει να γίνει. Ταυτόχρονα και με τι επιχειρήσει και με του ιδιώτες θα πρέπει να ασχοληθούμε. Μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή να αφιερώσει χρόνο στο θέμα το φορολογικό φορολογικό ε, και να δούμε ότι πρέπει να, ε, να εξετάσουμε, υπάρχουν και κείμενα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε κάθε διαφόρους τομείς και χαιρετίζουμε την ανακοίνωση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έργο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο που αναφέρθηκε από τον κύριο Πιτέλα σημαντικό θέμα που αφορούν το ποινικό θέμα, το ξέπλυμα χρήματο κλπ. Και γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθούν άλλε επιτροπέ όπω είναι η Νομική και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Δεν θα πρέπει να αρκεστούμε να γράφουμε διάφορα έγγραφα. Είναι το θέμα τη εφαρμογή του ελέγχου και των ενδεχομένων κυρώσεων κατά των προσώπων που δεν σέβονται του κανόνε. Όλα αυτά θα πρέπει να αναλυθούν ενδελεχώ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ψηφίσαμε στην έκθεσή μου μια έκθεση πρωτοβουλία για το ρόλο μας ε, μία από τις θέμες αξίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα ήταν να πολεμήσει για την εφαρμογή των ε, ε, κυρώσεων. Είμαστε υπέρ της τάξης σε παγκόσμιο επίπεδο που θα πρέπει να βληθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε στη διάθεσή σα, στη διάθεση τη Προεδρία και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σα βοηθήσουμε. Είναι σοβαρό θέμα και δεν θα εξαφανιστεί σύντομα από τι οθόνε των ραντάρ μα. Σα ευχαριστούμε κύριε και τώρα το λόγο έχει για την ο κύριο Δεμάζη. Κύριε Πρόεδρε, στο Panama Links το θέμα είναι εργονομένο έγκλημα των πλούσιων και των δυνατών. Η Mossack Fonseca με την εντολή τη ε, Deutsche Bank ξέπλυνε βρώμικο χρήμα και βοήθησε τη φοροδιαφυγή. Οι τράπεζε του Ισλαμικού κράτου ε, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το διεθνέ σύστημα SWIFT και έτσι με το χρή... βρώμικο χρήμα χρηματοδοτήθηκαν οι επιθέσει στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Πολύ μεγάλη και ευγενή αυτή η ελίτ στην λίστα της, του Παναμά. Ε, έχουμε λοιπόν τον ε, Ρώσους προαγωγούς, ε, Ουκρανούς, τον Ουκρανό Ολιγάρχη και Πρόεδρο Προσέσκο, τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κάμερον, FIFA, την σύζυγο του Κανιέτε και το Front National. Εγώ έχω το όνομά μου στο χρηματοκιβώτιό μου, στο χρηματοκιβώτιό μου και η πλειοψηφία του κόσμου αυτό κάνει. Για κάθε κεφρολογείται. Αυτό που ισχύει όμως είναι ότι η... αν η πλούσια θέλει μεγαλύτερα μερίδα της πίτας, αυτό υπονομεύει τους άλλους. Η συζήτηση για τον Παναμά όμως αποκαλύπτει και μια μεγάλη υποκρισία. Η Γερμανία ε, αντιστέκεται σε ένα δημόσιο μητρό των κατόχων τέτοιων πλασματικών εταιριών. Οι τράπεζες στη Γερμανία δεν φοβούνται τίποτα σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Οι Ολλανδοί δεν, δεν ε, φορολογούν ε, του φορολογικού παραδείσους, τα χρήματα που φεύγουν στου φορολογικού παραδείσους και οι ΙΠΑ έχουν την Delaware και μποκοτάρουν την ανταλλαγή απόψεων. Τι θα γίνει, όλοι θα μπουν σε μαύρη λίστα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ένα φορολογικό δίκαιο για τι ε, τράπεζες, ε, για τι εταιρείε. Χρειαζόμαστε ένα δημόσιο μητρό για τους πραγματικούς κατόχους πλασματικών εταιρείων. Χρειαζόμαστε ένα μητρό περιουσιών και χρειαζόμαστε και ένα τέτοιο μοντέλο για κάθε χώρα, όχι μαύρε λίστε και ανοησία. Αυτό που ζητάμε είναι μια μόνιμη εξεταστική επιτροπή για του ορολογικού παραδείσου Η πλειοψηφία εδώ πέρα στο κοινοβούλιο μετά το LuxLeaks θα έπρεπε να έχουν επιστρέψει στι πατρίδε του για να κοιτάξουν τι γίνεται. Γιατί το είχε πει και ο Ισού, άλλωστε ευκολότερο να περάσει καμίλα μέσα από το τρίπο μια βελόνα παρά να μπει πλούσιο στη βασιλεία του Θεού. Και πού να ξέρει ότι θα υπήρχε αμφρολογική παράδοση. Και παρόλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουμε αυτού του. Ε, φορολογικού παραδείσους αντί να κάνουμε ωραίε και ομορφε ομιλίες. Ο Πρόεδρος, για τους πράσινους το λόγο έχει ο κύριος Λαμπέρτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι πολίτες μας θεωρούν ότι δεν ε, λειτουργούν οι δημοκρατίες και ότι ωφελούνται οι λίγοι και αυξάνονται αυτοί που το πιστεύουν. Δέκα ημέρες μετά το σκάνδαλο των Panama Papers ε, η έγκριση μεθαύριο μια οδηγία που προστατεύει ή τέλο πάντων με πρόσχημα ότι προστατεύει ε, το επιχειρηματικό απόρριτο ε, θα, ε, θα κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά των δημοσιογράφων που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του Παναμά και τα Lux Leaks είναι σκάνδαλο και είναι επίθεση κατά τη δημοκρατία. απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω στον Επίτροπο Μοσκοβισή. πιο πριν τα λέγατε πιο χιουμοριστικά και πιο ελαφριά. Εγώ πρέπει να σα πω όμω ότι πλέον έχω απελπιστεί κύριε Μοσκοβίση. Τρία χρόνια ε, που αποκαλύφθηκαν τα Lux Leaks ε, και 16 μήνες έχουμε το reporting καναχώρα. Είναι υποχρέωση για κάθε τράπεζα χωρίς διάκριση μεταξύ των χωρών. Αλλά όλο αυτό τον καιρό ε, καθυστερείτε εσείς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθυστερείτε το reporting αναχώρα για όλες τις επιχειρήσεις και για όλες τις χώρες, γιατί δεν το θέλετε και λυπάμαι, συγγνώμη, δεν έχετε κανένα επιχείρημα, κανένα επιχείρημα βάσιμο και εύλογο για να καθυστερείτε τις εκθέσεις αναχώρα, το reporting αναχώρα. Κανένα επιχείρημα, μία ΜΜΕ που δρά μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας, ξέρει πόσους υπαλλήλους έχει στη Γαλλία και στο Βέλγιο, τι πόρου πληρώνει στη Γαλλία και στο Βέλγιο, τι τζίρο κάνει στη Γαλλία, τι τζίρο κάνει στο Βέλγιο. Μην έρχεστε να μου πείτε ε, ότι δεν το ξέρει, διότι τότε δεν είναι μια σωστή επιχείρηση και μικρέ επιχειρήσει μπορούν να σα δώσουν αυτά τα στοιχεία. Επίση, σε καμία χώρα, δεν, ε, καμία χώρα δεν υπάρχει στην οποία να μην μπορούμε να υποχρεώσουμε σε αυτή την ε, έκθεση αναχώρα. Άρα, μην μου λέτε καθυστερείτε, και η Business Europe ε, που εκπροσωπεί το ΜΕΝΤΕΦ και όλες τις ε, ομοσπονδίες και ενός επιχειρήσεων είναι αυτή που δεν το θέλει γιατί τη διαφάνεια θα την πληρώσουν ε, σε ό,τι αφορά τη φήμη τους όλες οι επιχειρήσεις. Εσείς συγγνώμη, αλλά αυτό που κάνετε είναι να προσπαθά να προστατεύσετε την καλή φήμη των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ο Γούλφ από το EFTD. Uh, thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά τη δημοσίευση των εγγράφων του Πανάμα έχουμε τη συνήθεια κατακραυγή από του πολιτικού που λένε ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν του φόρους που του αναλογούν Όπω και ο κ. Μοσκοβισή εδώ στην ομιλία του πριν από σήμερα. Θέλει οι πλούσιοι να πληρώσουν αυτά που του αναλογούν. Κύριε Μοσκοβισή, είσαστε ένα από του πλούσιου αυτού. Πάνω από 20.000 βγάζετε το μήνα. Έχετε άδεια διαμονή σε 3.000 το μήνα. Ε, επιδόματα, 6.000, ε, πράγματα τα οποία άλλος κόσμος μόνο ονειρεύεται. Είπατε ότι η διαφάνεια θα πρέπει να ισχύει για όλους. Και σας ρωτώ λοιπόν, θα συμφωνήσετε και εσείς και όλοι οι άλλοι επίτροποι να βάλετε δημόσια στο διαδίκτυο τις φορολογικές σας δηλώσεις για να δούνε την διαφάνεια στα φορολογικά των επιτρόπων ο κόσμος. Είπατε επίσης ότι θέλετε να καταπολεμήσετε τις φορολογικούς παραδείσους. Συμφωνώ. Θα καταπολεμήσετε λοιπόν το μεγαλύτερο φορολογικό παράδεισό σας, ε, τις Βρυξέλλε. Οι πιο πολλοί στον κόσμο στις στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλε πληρώνουν 45%. Εσείς, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι επιτροποί, πληρώνετε μέχρι και 8% μόνο φόρο ενώ σε όλες ε, τις άλλες χώρες ε, έχουμε 30-40-50% εσείς ε, απολαμβάνετε την πολυτέλεια των υψηλών μισθώσεων. Και οι, Ευρωπαί... και οι Ευρωβουλευτές πληρώνουν αυτά που αναλογούν στις χώρες σας. Οι Ευρωκράτες λοιπόν δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτε. Να λοιπόν που είναι το σκάνδαλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βούλφ. Ο κύριος Μόνο από το ENF. Κύριε Επίτροπε, έχουμε το νέο φορολογικό σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά που δεν είναι κάτι καινούριο το εθνικό μέτωπο, υπενθύμησε αποφασιστικότητα την οντολογική την πολιτική. Από τι αρχέ τη θητεία ψηφίσαμε όλα τα ευρωπαϊκά κείμενα για την καταπολέμηση τη απάτη, κατά τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή και τη βελτιστοποίηση. Επαληθεύστε το. Αντίθετα από τον κύριο Γιούνκερ, αρνούμεθα τη διτή γλώσσα και την υποκρισία κάποιων κυβερνήσεων. Οι φόροι που ξεφεύγουν από τα κράτη και τα κοινωνικά συστήματα θα πρέπει να τα πληρώσουν οι πολίτε, ενώ τα δημόσια ελλείμματα, τα οποία υποπτεύεται κύριε Μοσκοβιτσί, είναι στο ύψιστο σημείο. Είναι είναι ανισότητα ε, φορολογική που είναι ένα κρίμα κατά των λαών. Θα πρέπει να καταδικαστούν οι πολυεθνικέ που χρησιμοποιούν το σύστημα τη κυρίως κυρίω επιχειρήσει αμερικανικέ, το Google, το Apple και το Facebook, το Starbucks κλπ. Το αθέμα τους είναι να ξεφεύγουν από τη φορολόγησή τους μέσω αμφισβητουμένων ε, πρακτικών. Θα πρέπει όμως ε, και να βρούμε και ποιοι είναι και οι διάφοροι οι λογιστές, οι δικηγόροι, οι HCBS, οι διάφορες τράπεζες, UPS κλπ. Πέρα από τις απλές καταδίκες της αρχής της ε, απάτης, λείπει η έρευνα η σωστή που πρέπει να γίνει. Δεν έγιναν αποκαλύψει για του Αμερικανού φορολογικού παραδείσου. Καμία προσωπικότητα από τη Βόρεια Αμερική, καμία μεγάλη τράπεζα τη Wall Street α, κάνει κερδοσκοπία. Διότι ξέρουν ότι εκείνοι που χρηματοδοτούν είναι ιδρύματα που είναι το Ford, και Kennedy, η Rockefeller, η Kellogg και κάποιο κύριο όρο. Όταν ξέρουν ποιοι κρύβονται από εκεί, ξέρουμε από πού υπάρχει η διαφυγή και ποιοι το εκμεταλλεύονται. Στον παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο σήμερα είναι ένα στόχος αυτός που έχουν ε, και ακολουθούν επιχειρήσεις. Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Μονό. Μπλε κάρτα. Από τον κύριο Λαύρη. Ναι κυρία Πρόεδρε, δυόμιση λεπτά ακούσαμε ε, τον κύριο από το, λαϊκό, από το ε, εθνικό μέτωπο, αλλά να μην ε, μιλάει ουσιαστικά για έναν λογαριασμό στον Παναμά. Η βασική εταιρεία που ε, έκανε τις επικοινωνίες, ανέλαβε την επικοινωνία της προεκλογικής εκστρατείας του εθνικού μετώπου ήταν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, μέσα σε αυτά τα έγγραφα. Μήπως θα έπρεπε να έχει εκμεταλλευτεί 2,5 λεπτά για αυτοκριτική ο κ. Μονό. Ωραία τα είναι η απάντηση. Αλλά ξέρετε, εμεί καμία σχέση δεν έχουμε με αυτέ τι ε, υποθέσει φορολογικών παράδεισων. Εγώ μιλάω για το εθνικό μέτωπο, έτσι, εντάξει. Εσείς αναφερθήκατε σε δύο άτομα ουσιαστικά που είπαν όμως ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Εντάξει, Εντάξει, υπάρχει διαφάνεια, είναι τα πάντα δεδηλωμένα. Ο κύριο Λεπέν δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, άρα πρόκειται για συκοφατική δυσφήμιση. Στηρίζεστε, βασίζεστε πίσω από το, πώ να το πω, από το. Από το... Κόβετε το μικρόφωνο. Σα ευχαριστώ, συνάδελφοι. Σα παρακαλώ λίγη ησυχία, γιατί αυτή είναι μία από τι απόψει. Και ο έχει το Οι πρόσφατε αποκαλύψει σχετικά με τι υπεράκτιε εταιρείε στον Παναμά απλά επιβεβαίωσαν τα όσα ήδη γνωρίζαμε ή έστω υποψιαζόμασταν. η πολιτική τάξη της ευρώπης ακολουθεί κατά πόδα στο παράδειγμα των διεφθαρμένων επιχειρηματιών. πολλοί εκπρόσωποι και των δύο αυτών τάξεων θεωρούν πως είναι υπεράνω του νόμου την ίδια στιγμή που επιβάλλουν στους πολίτες μέτρα άγριας λιτότητας και εμφανίζονται ως σταυροφόροι ενάντια στη φοροδιαφυγή. πόσα από αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί πόσα προέρχονται από παράνομε δραστηριότητε και πόσα είναι νόμιμα; υπάρχει σοβαρότατο ηθικό ζήτημα και πρέπει όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση να λογοδοτήσουν και να αναλάβουν τι βαρύτατε ευθύνε του. θα πρέπει να αναλάβουμε δράση για την ανακάλυψη όλων όσων διατηρούν λογαριασμού σε υπεράκτιε εταιρείε καθώ τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει είναι ένα ελάχιστο κλάσμα μπροστά στο συνολικό αριθμό. το σημαντικότερο όμω είναι να πάρουμε μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν την επανάληψη του φαινομένου. οι υπεράκτιες εταιρείε δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό πέρα από το να διευκολύνουν του έχοντες ώστε να αποφεύγουν τα βάρη που του αναλογούν πρέπει να επανεξετάσουμε το καθεστώς τους σε ολόκληρη την ευρώπη. εξυπηρετεί πράγματι την κοινωνία η ύπαρξή τους; υπάρχει έστω μια αληθοφανής δικαιολογία για τη λειτουργία τους; επειδή η απάντηση είναι πως στην ουσία δεν υπάρχει καμία πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση της πλήρους απαγόρευσης δραστηριοποίησης υπεράκτιων εταιριών. οποιαδήποτε εταιρεία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην ευρώπη θα πρέπει να αποκτά φορολογική έδρα εντό τη ένωση φυσικά εταιρείε φαντάσματα χωρί κανένα αντικείμενο λειτουργία δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. όμω φοβάμαι πω δεν υπάρχει πολιτική βούληση για τέτοιου είδου μέτρα γιατί πιθανότατα όπω αποκαλύφθηκε πρόσφατα μεγάλο μέρο των εταιρεών αυτών ανήκει σε πολιτικού. Την εξή ερώτηση είχα να σα θέσω. Δεν πιστεύετε ότι αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, μάλλον ε, καταλυστεύει του Ευρωπαίου πολίτε 80 δις αναμήνα, αυτό ουσιαστικά είναι όπω ο το δασόν, ότι τελικά θα ξαναδίνει στον κόσμο. Τα αυτά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ε, η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα καταλυστεύει τους ευρωπαίους πολίτες και παράλληλα όπως αποδείχθηκε από τα panama papers πολιτικοί έχουν βάλει πάρα πολλά χρήματα μαύρα σε αυτές τις υπεράκτιες εταιρείες. Επόμενοι α, ομιλητές, ο κύριος Νίντερμαϊερ. Μάιερ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το σκάνδαλο των γράφων του Παναμά δείχνει ότι θα πρέπει να είμαστε τολμηροί και αποτελεσματικοί για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της φορολογήσεως. Ο λόγος δεν είναι μόνο ότι πρέπει να συλλέγονται τα χρήματα αυτά για τον προπολογισμό, αλλά είναι και θέμα αξιοπιστίας των κυβερνήσεων και τη δικαιοσύνη στην αγορά. Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εγγράφων του Παναμά και των LuxLeaks. Στα έγγραφα του Παναμά ασχολούμεθα περισσότερο με άτομα και όχι με επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι στα έγγραφα του Παναμά βλέπουμε περισσότερο φοροδιαφυγή και όχι φοροαποφυγή και οι πηγές των χρημάτων όσον αφορά του λογαριασμού του Παναμά δεν είναι ξεκάθαροι. Θα πρέπει να σημειώσουμε σε πολλέ περιπτώσεις τα έγγραφα του Παναμά ε, έχουμε παλιές περιπτώσεις το λέω αυτό διότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τομέα της χειραγώγησης, της φορολόγησης. Αυτά που περιγράφονται στα έγγραφα του Παναμά μιλάνε για θέματα για τα οποία υπήρξε δράση τελευταία, όπως αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και βελτίωση της καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος. Γι' αυτό καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια αναθεώρηση, να δει κατά πόσο τα μέτρα που εθετήθηκαν αρκούν και ενδεχομένω ποια είναι τα κενά, ποια στοιχεία λείπουν από τον κανονισμό που ασχολούνται με τα προβλήματα περιγράφοντα τα έγγραφα του Παναμά. Επίση, θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει ε, στο πρόγραμμά τη για τη φορολόγηση, κυρίω τη φορολόγηση των εταιριών και τη βελτίωση τη συλλογή ε, του ΦΠΑ. Έχετε την πλήρη υποστήριξή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αποκαλύψεις ε, των εγγράφων του Παναμά. Πρώτα απ' όλα ε, μας επιβάλλουν να γνωρίσουμε την καταπληκτική δουλειά ε, αυτών των δημοσιογράφων αλλά βέβαια να ευχαριστήσουμε πρέπει και τους καταγγέλλοντες που έδωσαν αυτά τα στοιχεία. Ξέρετε ότι ένας από αυτούς που απεκάλυψε το LuxLeaks ε, θα δικαστεί για αποκάλυψη επιχειρηματικών ε, μυστικών και εμπορικών μυστικών. Ε, συμφωνώ με το εγκόμιο που έπλεξε ο Επίτροπος Μοσκοβίσης στους δημοσιογράφους, όμως έχουμε αυτούς που καταγγέλουν και οι οποίοι διώκονται δικαστικά, ενώ έχουν κάνει τόσο καλό. Τώρα, ε, αυτό που βλέπουμε με τα έγγραφα του Παναμά είναι το, ε, η κορυφή του παγόβουνου μόνο. Το θέμα είναι τι ε, είναι η φορολογική παράδοση. Πρέπει να οριστούν με σαφή διαφανή κριτήρια και ποιοι συνεργάζονται με αυτούς. τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλω να ασκήσω κριτική γιατί σας εγκομιάζω και σας ενθαρρύνω. το Συμβούλιο όμως δεσμεύεται να είναι πιο αποφασιστικό. Τι έκανε τελικά όμως το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τη φορολογία, τίποτα, μηδέν. Υπάρχει εμπλοκή, υπάρχει απάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν κουνιέται το Συμβούλιο, βήμα, ρούπι, αυτό είναι αδράνεια. Σας ευχαριστώ πολύ και επόμενος ομιλητής είναι ο κύριο Λούνας. Ένα λεπτό, ναι. Κυρία Πρόεδρε, αντισόπιτα έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα σκάνδαλα του Παναμά. Ε, γιατί πολύ απλά δεν θέλουν κάποιοι να συμβάλλουν και προδιαφεύγουν ένα κοσμάκι τελικά πληρώνει του τους φόρους και αυτό προφανώς δεν μπορεί να το επιτρέψουμε. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εφοριών και αν ε, δεθεί ε, ερώτημα και ζήτημα για να τη σύσταση μόνιμη επιτροπή, θα υποστηρίξει το ΕΝΒΑ. Να υπάρχουν δηλαδή ε, ομόνια συνεργασία και όχι διαρκή φοροαποφυγή γιατί ιδάλω ε, αυτό που ισχύει για τον... η πραγματικότητα είναι ότι στον ιδιωτικό κλάδο συχνά τρία τέταρτα δίνονται από τα έσοδα στι αρχέ. και έτσι ε, αυξάνονται διαρκώ τα χρέη και κανείς φυσικά δεν μπορεί να θέλει να δανείσει σε ε, άρρωστε κυβερνήσει και έτσι λοιπόν ε, αναγκάζεται συνεχώ να χτυπώνει περαιτέρω χρήματα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συνάδελφοι, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Αν θέλουμε να υπάρχει δίκαιη κατανομή των ε, φόρων, θα πρέπει ο καθένας να συνδράμει αυτή την αναλογία, ακόμα και αυτοί που προτιμούν να είναι κατά από στον Παναμά. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι η υπόθεση εδώ πέρα του Παναμά είναι η μεγαλύτερη της ιστορίας με 11,5 εκατομμύρια έγγραφα και έχουμε μια φοβερή κατάσταση. Είναι ξέραμε ότι υπήρχαν φορολογική παράδειση αλλά οι διαστάσεις είναι τεράστιες και μιλάμε για πρόσωπα της παγκόσμιας ελίτ, όχι μόνο επιχειρηματίες, ε, σκηνοθέτες, ε, καλλιτέχνες και βεβαίως πολιτικοί και υπάρχει άρα η εντύπωση στον πολίτη ότι δεν αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά το ζήτημα γιατί μπλέκονται πολιτικοί. Έτσι υποβαθμίζεται η δημοκρατική νομοποίηση. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το, η πρώτη επιτροπή ήδη έχει βάλει τις βάσεις. Δεν ήμασταν τυφλοί απέναντι στο ζήτημα. Ζητήσαμε τα αναγκαία μέτρα, ζητήσαμε από την Κομισιόν να υποβάλει κάποιες προτάσεις και ορισμούς. Χρειάζεται όμως μια επιτροπή τάξη η οποία θα έχει πραγματικά αρμοδιότητες να διερευνήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ματίας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε αν τα έγγραφα αυτά είναι απλά η κορφή του παγόβουνου θα έλεγα πως ε, θα έπρεπε να μιλάμε για εμάς τους ιδίους ε, και για την ύπαρξη φορολογικών παραδείσων. Σε κανένα δεν αρέσουν οι φορολογικοί παραδείσοι, αλλά κανένας δεν κάνει και τίποτα. Οπότε, για να υπάρχει φορολογική εναρμόνιση, πρέπει να φροντίσουμε οι μικρομεσαίες εταιρείες να μην αναγκάζονται και να προσπαθούν να αποφύγουν τη φορολογία. Υπάρχουν χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μαδέιρα που λειτουργούν ε, ως ε, φορολογική παραδείσοι. Και επειδή έχουμε τόσους φορολογικούς ε, παραδείσου είναι σοβαρό το πρόβλημα. Το γεγονό, λοιπόν κύριε Μοσκοβισή ότι έχουμε φορολογικού παραδείσου εντό τη Ευρώπη σημαίνει πως θέλουμε ένα μήνυμα προ πολίτε. ότι ε, αν ε, φοροδιαφεύγει 100 ευρώ είσαι εγκληματία, αν διαφοροδιαφεύγεις 100.000 είσαι επιχειρηματία. Ε, ο κύριο Γκίγκολτ συνάδελφοι επίτροποι το σκάνδαλο αυτό δεν είναι κυρίως φορολογικό, είναι σκάνδαλο ξεπλήματος χρήματος με φορολογικές πτυχές. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές ήδη παραβιάζουν ε, όσον αφορά την Ευρώπη την υφιστάμενη νομοθεσία περί ξεπλήματος χρήματος που ισχύει από το 2005. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Εμένα με ενημέρωσε ένας πληροφοριοδότης που ήταν σε επαφή με την Κομισιόν εδώ και χρόνια για να επιμείνω στο ότι δεν εφαρμόζεται η υφιστάμενη νομοθεσία στην πράξη. Και άρα πρέπει το Κοινοβούλιο να ερευνήσει γιατί τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί η Κομισιόν δεν επιμένει ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Οπότε, ζητάω από την Κομισιόν να ξεκινήσει σε παραβάση κατά των κρατών μελών ε, για να εφαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία. Και το Κοινοβούλιο αυτό πρέπει να ξεκινήσει μια διερευνητική, μια εξεταστική επιτροπή για να δει το θέμα της μη εφαρμογής. Τέλος, είναι σημαντικό αν ξεκινήσει η νέα επιτροπή, να μην μπει στο σιρτάρι η δουλειά που έχει γίνει στην πρώτη επιτροπή τάξε, γιατί οι πολίτες δεν θα δεχτούν να πηγαίνουμε από το ένα σκάνδαλο στο άλλο και να μην τελειώνουμε ποτέ τίποτα. Είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΣΑ, χάνονται από τους εθνικούς προπολογισμούς γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων. Λοιπόν αυτό να είναι πρώτη προτεραιότητα. Αν δεν ήταν θα έπρεπε να γίνει μετά τα Panama Papers. Και θα πρέπει λοιπόν τα κέρδη να φορολογούνται εκεί όπου υπάρχει φορολογική δραστηριότητα. Έχουμε λοιπόν αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με το πρόγραμμα των 15 σημείων όσον αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων με το κλείσιμο των ε, παραθύρων που υπάρχουν. Ήδη 96 χώρες έχουν συμφωνήσει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Ο Παναμάς δεν το κάνει, οι ΙΠΑ δεν το κάνουν και ξέρετε πως το Delaware έχει περισσότερες εταιρίες από ότι ανθρώπους, κατοίκους. Και ξέρετε πως χρειάζεται ένα email και η εταιρεία σου έχει ιδρυθεί. Επίσης ε, σημαντική είναι και η έκθεση που βρίσκεται τώρα στην Αρμόδια Επιτροπή και οι αναφορές αναχώρα για τις επιχειρήσεις που έχουν τζίρο πάνω από κάποια εκατομμύρια ευρώ. Αυτά όμως δεν επαρκούν. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και χρειάζεται μια παγκόσμια δικτύωση, ένα παγκόσμιο αρχείο των φορολογουμένων και να υπάρξει και μια αυστηροποίηση των προθεσμιών παραγραφής. Ευχαριστώ. κύριο Κάζα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές έτσι ώστε να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Δυστυχώς όμως τα Panama Papers δείχνουν ότι αυτοί που έχουν αρκετή εξουσία και οικονομικά μέσα μπορούν να παρακάμψουν τους κανόνες και μπορούν να αποκρύψουν <clears throat> κεφάλαια μέσω περίπλοκων ε, κατασκευών θα έλεγα και αρχιτεκτονικών. Η Μάλτα έχει αυστηρότατους κανόνες συμβατούς με τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Έχουμε μια δικαιοδοσία υψηλού επίπεδου και με αυστηρότατες ε, ρυθμίσεις και κυρώσεις. Οι δράσεις της μικρής κλίκας που ήταν στην εξουσία προσέφυγαν λοιπόν αυτοί στις υπηρεσίες των εταιριών του Παναμά αλλά δεν αντιπροσωπεύουν τη Μάλτα, δεν αντιπροσωπεύουν την πειθαρχία και την τιμιότητα των κατοίκων της Μάλτας οι κάτοικοι της Μάλτας μαζί με σας, μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου καταδικάζουν αυτές τις πράξεις διαφθοράς. <clears throat> Τέτοιου είδους καταστάσεις δεν θα γίνουν ανεκτές στο μέλλον. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τα μέλη του Κοινοβουλίου και από την όλη πλευρά που μίλησαν και που εκπροσωπούν τη χώρα μου. Η Μάλτα θα πρέπει επειδή είναι ειλικρινής να παραμείνει στα υψηλά ευρωπαϊκά επίπεδα. Από τον κύριο Κουκάν μπλε κάρτα. Κύριε Κούκαν έχετε το λόγο. Πρόεδρε, μία ερώτηση άμεση στον κύριο Κάσα. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε, είναι αλήθεια ότι θα υπάρξει μία ψήφος εμπιστοσύνης στην Μάλτα λόγω ακριβώς των Panama Papers. Απλή ερώτηση, απλή απάντηση. Βεβαίως, Πρόεδρε, επιβεβαιώνω ότι η αντιπολίτευση ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης, έλεγχο της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Βέβαια δεν ενδιαφέρονται ε, για τα Panama Papers, ενδιαφέρονται για νέες εκλογές είναι ε, νομίζω απαραίτητο οι υπεύθυνοι για αυτό το σκάνδαλο να παραιτηθούν. Θυμίζω ότι χιλιάδες κάτοικοι της Μάλτας από όλε τις κοινωνικές κατηγορίες πήραν μέρος στις διαμαρτυρίες. Δυστυχώς υπάρχει μια ενορχιστρωμένη επίθεση εναντίον αυτών που πήραν μέρος σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι τίμοι, που έχουν κάνει πολλά καλά στη χώρα τους. Είναι ένα σκάνδαλο λοιπόν για την κυβέρνηση που επιτρέπει τέτοιες ε, επιθέσεις. Σας ευχαριστώ. Κύριο Σίμων είναι ο επόμενος ομιλητής. Ένα λεπτό έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, τον τελευταίο χρόνιο στην Ευρώπη για αυτά τα ζητήματα έχουμε κάνει περισσότερα πράγματα από τα προηγούμενα χρόνια γιατί είχαμε μια σύμπτωση του τύπου των ε, καταγγελόντων της Κομισιόν αλλά ιδιαίτερα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ειδική του επιτροπή την τάξε και την τάξε 2 που άσκησε δημόσια πίεση. Αν δούμε τώρα την εξαιρετική έρευνα της Deutsche Zeitung με τα Panama Papers και έχουμε μια νέα διάσταση όπου περνάμε σε μεμονωμένα άτομα, σε ομίλους, σε συλλόγους. Πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί αυτή η πίεση. Πρέπει να υπάρξει μία εξεταστική επιτροπή η οποία θα μας δώσει τα απαραίτητα μέσα σε συνεργασία με την Κομισιόν μακροπρόθεσμα να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη για να θελήσουν να περάσουν την απαραίτητη νομοθεσία σε συνεργασία μαζί μας για να κλείσουν τα παραθυράκια που υπάρχουν ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ρόνελερ, ναι, ένα ναι. λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το LuxLeaks, ε, LuxLeaks ε, και το σκάνδαλο του Παναμά τώρα. Τι άλλο θέλουμε για να σταματήσουμε πια με την ε, φόρα αποφυγή. Νομίζω ότι έχουμε αρκετέ πληροφορίε μέχρι τώρα, ξέρουμε αρκετά τι συμβαίνει. Αυτό που λείπει είναι βούληση από όλα τα πολιτικά κόμματα σε όλε τι χώρε. Τώρα ήρθε η ώρα να δράσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, είναι σαφέ ότι τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν και παγκόσμιε λύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί από μόνη τη να αποφύγει τέτοιε απάτε. Χρειάζεται διαφάνεια σε διεθνέ επίπεδο, από όλου δηλαδή. Ο υπουργό Σόμπλερ, για παράδειγμα, στην Γερμανία. Και αυτός πρέπει να βοηθήσει. Οι λύσεις δεν πρέπει να είναι μόνο οικονομικές. Οι προνομιούχοι έτσι κι πάντα τα καταφέρνουν και ξεφεύγουν. Και αυτό που κάνουν είναι ότι πλήττουν την ηθική πτυχή των πραγμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν φορολογικές πληροφορίες και να καταπολεμηθούν όλοι οι φορολογικοί παράδοση με κάθε τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής Βιέγας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο παραπάνω που μας υπενθυμίζει μια πραγματικότητα που δεν είναι καινούρια. Είτε πρόκειται για τα LuxLeaks είτε για άλλα τέτοια σκάνδαλα, τώρα φτάνουμε και στα σκάνδαλα του Παναμά. Πρόκειται για μια απορρίθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που άρχισε ήδη από τη δεκαετία του 70. Έχουμε και την ιδιωτικοποίηση πολλές φορές των δημοσιονομικών. Όλα αυτά έχουν αρχίσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για διαρθρωτική κρίση, η οποία απαιτεί μέτρα ουσίας για να αντιμετωπιστούν η φορολογική παράδεισοι και να καταπολεμηθούν οι κάθε είδου φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε την φοροαποφυγή και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις φορολογικές πληροφορίες. Να μην βρίσκουμε εμπόδια σε αυτά. Κάτι πρέπει να δείξουμε ότι κάνουμε για να μην συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. σε ευχαριστούμε. Μπλε κάρτα για σας. Ή προτιμάτε να περάσετε στο Catch the Eye. Οι αποκαλύψεις, λέει η κυρία Ζόλη, της προηγούμενης εβδομάδας, δεν σας έχω δώσει ακόμα το λόγο, περιμένετε. Ναι, εγώ προτιμάω Catch the Eye τότε, αντί για μπλε κάρτα. Καλώς, τότε συνεχίζουμε. Η κυρία Ζολή έχει το λόγο. Παρακαλώ, κυρία Ζολή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ωραία, αρχίζω λοιπόν και πάλι και το χρόνο. Λοιπόν, κύριε Πίτροπε, οι αποκαλύψεις της προηγούμενης εβδομάδας μας υπενθυμίζουν ένα πράγμα, ότι οι κανόνες για την νομιμοποίηση και για την αποφυγή νομοποίησης παράνομου χρήματος δεν τηρούνται. Με διάφορα κόλπα. Ούτε οι χώρες μέλη τηρούν τους κανονισμούς, ούτε σε διεθνές επίπεδο γίνεται ο κατάλληλος έλεγχος η νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος έχει γίνει μια επιχείρηση σαν οποιαδήποτε άλλη. Και έχουμε φτάσει σε επίπεδα παροξισμού. Οι κυβερνήσεις μας έχουν διπλό λόγο. Και όλα αυτά έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κόσμου τα μυστικά και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές που προσπαθούν να ερευνήσουν τέτοια σκάνδαλα μας έχουν αποκαρδιώσει όλους. Δεν καταφέρουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός που φταίει, πώς γίνονται οι απάτες και πώς θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Πρέπει να ρίξουμε λίγο φως στις απάτες αυτές. Σε μεγάλη κλίμακα. Γι' αυτό και η ομάδα μου πρότεινε να δημιουργηθεί μια ερευνητική επιτροπή. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους που μας υποστήριξαν στο έτοιμά μα αυτό. Κύριε Επίτροπε, δεν θα αφήσουμε τα σκάνδαλα να ακολουθούν το ένα το άλλο χωρίς να κάνουμε τίποτα. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί, πώς είναι δυνατόν, ενώ εσείς μπορείτε να κάνετε πολλά εφόσον σας στηρίζει ο κόσμος, δεν μας προτείνετε ένα πραγματικό μέτρο. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής. Μπαγέ, μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ο συγγραφέας Μωρά τον προηγούμενο αιώνα το έλεγε αυτό και αυτό έρχεται στο μυαλό μου όταν ε, σκέφτομαι τη δουλειά που έκανε αυτή η σύμπραξη δημοσιογράφων και αποκάλυψε το σκάνδαλο του Παναμά. Και αυτό έρχεται στο μυαλό μου όταν ε, διαπιστώνω τα στατιστικά στοιχεία που βγαίνουν από τις έρευνες οι σοσιαλιστές και άλλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και ζητήσαμε μια ερευνητική επιτροπή και ελπίζω να υπάρξει πλειοψηφία υπέρ της δημιουργίας μιας τέτοιας επιτροπής. Γιατί μετά από το LuxLeaks έγινε κάτι τέτοιο. Ξέρετε, τα μέλη βέβαια της επιτροπής αυτής βρέθηκαν στο ωριά τους. Υπήρξε και απειλή για να μας δώσουν τα συμπεράσματά τους. Πρέπει όμως να το κάνουν. Βέβαια παρόλα αυτά τελικά καταλήξαμε σε πολλές φιλόδοξες προτάσεις οι οποίες δυστυχώς δεν εισακούστηκαν από τις 28 χώρες μέλη και το είπατε και εσείς κύριε Επίτροπε. Γι' αυτό και ζητάω Όντω, να δημιουργηθεί αυτή η Ερευνητική Επιτροπή. Είναι ο μόνο τρόπο για να ερευνήσουμε σε βάθο το νέο αυτό σκάνδαλο και να αποδώσουμε ευθύνε στου υπεύθυνου και να εγκαθιδρύσουμε του σωστού οργανισμού. Και να διευρύνουμε την περίμετρο τη έρευνά μα ώστε να αντιμετωπίσουμε του μηχανισμού νομοποίηση του παράνομου χρήματο που είναι διεθνεί και το γνωρίζουμε όλοι. Οι επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει επιτέλου να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο οι πολίτε που πρέπει να σφίγγουν τη ζώνη, ότι Υπάρχουν χρήματα, απλώς πρέπει να έχουμε το θάρρος να πάμε και να τα βρούμε εκεί που υπάρχουν. Πρόεδρος Μόνικα Μακοβέη είναι επόμενη ομιλήτρια. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Μακοβέη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το σκάνδαλο που ξέσπασε τα Panama Papers είναι τρομερό, χωρίς προηγούμενο. Δείχνει ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου ολίγοι πλούσιοι, ολίγοι ισχυροί καθοδηγούν τα πάντα και οι υπόλοιποι, η μεγάλη πλειοψηφία, εργάζονται, υδρώνουν και απλά πληρώνουν φόρους. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα λοιπόν στις χώρες μας λόγω ακριβώς των φορολογικών παραδείσων και το διαφυγόν κέρδος για τους εθνικούς προϋπολογισμούς μπορεί να φτάνει και τα 3 ε, ευρώ φυσικά είναι ένας αριθμός ο οποίος προκαλεί ήλιγκο, δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι αντιπροσωπεύει. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια εγκληματική οργάνωση από λίγους που μας κοροϊδεύουν και απλά κερδίζουν αφορολόγητα χρήματα προκαλούν τις οικονομικές κρίσεις, σκοτώνουν ουσιαστικά μέσω της συμπεριφορά τους, πολύ αυτοκτόνησαν λόγω της ανέχειας της οικονομικής ή και πολλοί έχασαν τη ζωή τους λόγω ακριβώς της φτώχειας τους. Urban κρέσπο, ένα λεπτό. Σεβαστείτε το χρόνο σας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο απασχολεί τις ευρωπαϊκές αρχές δεν είναι το μέγεθος της φορολογικής απάτης, το Panama Papers, αλλά το ότι θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των φοροφυγάδων. Φύγονται πολιτικοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι λέγουν ότι είναι πατριώτες αλλά κρατούν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Βλέπουμε τι κάνει και ο Επίτροπος Κανιέτε που μέσω των συγγενών του υπονομεύει για μια ακόμη φορά την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι μεγάλες περιουσίες στην Ευρώπη δεν θέλουν τον Παναμά. Παίρνουν το τρένο και πηγαίνουν στο Λουξεμβούργο, στην Ελβετία ή στην Ανδόρα. και οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες βοηθούν τους μεγάλους αυτούς ε, πελάτες σε συνεργασία με το γραφείο Μόσα Fonseca. Την ίδια ακριβώς εβδομάδα που συζητάμε το Panama Papers συζητιέται και μια οδηγία για τα εμπορικά εμπιστευτικά στοιχεία που προστατεύουν αυτούς τους ε, ε, πατεώνες. Αυτό λοιπόν δεν είναι ε, μια, ένα απλό φαινόμενο κρίσης, είναι μια μεγάλη απάτη. Σκοτ Κέιτο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή μέχρι στιγμής έχει εστιαστεί σε διεφθαρμένους πολιτικούς και ε, απλούς εγκληματίες ε, που έχουν κρύψει τα λεφτά τους εκεί πέρα αλλά βεβαίως σημασία έχει και το κύκλωμα που τους διευκολύνει μισές από τις ε, εταιρείες που εμφανίζονται εκεί πέρα 130.000 στο σύνολο έχουν έδρα στα British Virgin Islands. Ακριβώς η σχέση μεταξύ αυτών των υπεράκτιων επικρατιών και του City του Λονδίνου διευκολύνει τους πλουσίους. Ο David Cameron παρουσιάζεται ως υπέρμαχος της φορολογικής διαφάνειας, όμως προσωπικά παρενέβη για να εξασθενήσει διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος, ειδικά για καταπιστεύματα, τα οποία τώρα ξέρουμε ότι ε, ωφελήθηκε και ο ίδιος. Έχουμε λοιπόν αυτές τις ε, βρετανικές υπεράκτιες κτίσεις οι οποίες βρίσκονται σε ένα νομικό κενό οι οποίες μέσω της φοροδιαφυγής στερούν υπηρεσίες από τους ευπαθείς στην χώρα μου. Αυτά περί Κάμερον και όλοι στην ίδια βάρκα είμαστε. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κόφοντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα Panama Papers μας δείχνουν με ποιο τρόπο μια ελίτ διεφθαρμένη παίζει τα δισεκατομμύρια στους φορολογικούς παραδείσους. Αποφεύγουν την πληρωνή φόρων, ξεπλένουν χρήμα, χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και μιλάμε μόνο για την κορυφή του παγόβουνου. Ένα δικηγορικό γραφείο, μία χώρα, ενώ υπάρχουν τόσες πολλές. Το 8% των ιδιοκτησιών με τον ένα ή άλλο τρόπο κρύβονται σε αυτές τις χώρες. Δισεκατομμύρια φόρων που διαφεύγουν τους ευρωπαϊκούς, από τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς. Δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών, της υγείας, της εκπαίδευσης, και φυσικά στην Ευρώπη ε, η φορολογία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ ψηλότερη από ό,τι στις πολύ μεγάλες. Όλα αυτά δυστυχώς διαγράφουν την έννοια της εμπιστοσύνης στις οικονομίες μας. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στα λεγόμενα country by country reporting έτσι ώστε να ονοματίσουμε τους απαταιώνες, να ονοματίσουμε τις χώρες όπως ο Παναμάς και τα British Virgin Islands, και να ελέγξουμε όλες τις νομικές κατασκευές που χρησιμοποιούνται για τη φοροδιαφυγή όπως τα κασταπιστεύματα και τις επιχειρήσεις όπως τους, τους ε, Μόσα Φωσέκα που ε, διευκολύνουν αυτή την φοροδιαφυγή. Κύριος Μελανσόν. Από το 2005 έχουμε ένα σκάνδαλο το χρόνο όσον αφορά τα φορολογικά σκάνδαλα. Η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα, ότι όλα αυτά πια είναι στο γενετικό κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ευνοεί τις φορολογικές απάτες. Απαγορεύεται η αναρμόνιση φορολογική και το άρθρο 63 διευκολύνει όλες τις συναλλαγές και απαγορεύει να βάζουμε όριο αναχώρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράνομο τελικά και κλέξατε ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναν αναμειγμένο σε τέτοια φορολογικά σκάνδαλα και μετά από τόσες συνεδριάσεις στην Αρμόδια Ερευνητική Επιτροπή τίποτα δεν βρήκατε. Μετά όμως βγήκαν τα σκάνδαλα αυτά και αυτοί οι οποίοι τα έβγαλαν βρέθηκαν να διώκονται και να πρέπει να πληρώσουν πρόστιμα. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε, τώρα με το σκάνδαλο του Παναμά, πάλι τα ίδια θα έχουμε. Η Bank General, Γαλλική Τράπεζα, αυτή άνοιγε επιχειρήσει offshore. Ο πρόεδρό τη, κάτω από είπε ψέματα Ποιο διώκεται όμω εγώ, επειδή λέει δυσφήμισα. Τίποτα δεν κάνετε με τα νέτρα που παίρνετε. Και εγώ χτυπάω το κουδούνι του συναγερμού, το καμπανάκι του συναγερμού, γιατί όσοι λένε την αλήθεια διώκονται τελικά. Ευχαριστούμε Μαραγκάλ τώρα. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Παναμάς είναι η κορυφή του παγόβουνου. Κάποιοι λένε ότι κατά κάποιο τρόπο είναι με ένα ξεπερασμένο σύστημα. Ίσως, αλλά βλέπουμε ότι διάφορες ε, εταιρείες κρύβουν τα χρήματά τους σε τέτοιους φορολογικούς παραδείσους και χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκα συστήματα. Η Ερευνητική Επιτροπή που προτείνουμε θα έπρεπε να ερευνήσει ολόκληρο το θέμα, κάθε του διάσταση. Εδώ δεν πρόκειται μόνο για ένα ηθικό ζήτημα, πρόκειται για ισότητα αλλά και για οικονομική επάρκεια. Δεν πρέπει πια να έχουμε τέτοια κεφάλαια παράσιτα τα οποία πλήττουν την ευημερία μας, αλλά να προωθήσουμε τα παραγωγικά κεφάλαια. Την ευθύνη την έχουν οι υπουργοί, οι πρόεδροι κυβερνήσεων, πρωθυπουργοί, ένας ενεργομέλος ακόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτοί φταίνε. Καταδικάζουμε το σύστημα εκείνο το οποίο νομιμοποιεί αυτά τα συστήματα. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό αν δεν σιωπούσαμε. Εμείς σιωπούμε. Πότε θα αρχίσουμε λοιπόν να εφαρμόζουμε προληπτικά αλλά και διορθωτικά μέτρα που να είναι κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής. Χαρέκια Τόντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η φορολογική παράδοση, παράδεση μας κλέβουν, έτσι είπε ο κύριος Μοσκοβισή και έχει δίκιο. Μας κλέβουν όλους εμάς, τους πολίτες, ε, τα δημοσιονομικά των χωρών μελών, την ευημερία μας και νομιμοποιούν ε, μαύρο χρήμα, αλλά και το κλέβουν από τους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να ανακτήσουμε τα χρήματα αυτά και για να το κάνουμε αυτό έχουμε μπροστά μας μια καταπληκτική ευκαιρία. Καταγγέλουν οι πολίτες, είναι ανακτισμένοι και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τα πράγματα καλά, όχι βέβαια μέσω από μια καταστροφική προσέγγιση, όχι να τα αλλάξουμε όλα, να τα φέρουμε τα πάνω κάτω, αλλά σιγά σιγά να παίρνουμε μέτρα το χρόνο που μας χρειάζεται να το κάνουμε, αλλά να πρόκειται για μια πραγματική φορολογική επανάσταση στον κόσμο μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Ας αρχίσουμε να δούμε τι σημαίνει ακριβώς φορολογικός παράδεισος. Ας φτιάξουμε συνενετικά ένα κατάλογο των φορολογικών αυτών παραδείσων και ας πάρουμε μέτρα εναντίον τους. Ας συμφωνήσουμε με τις τράπεζες να μην πηγαίνουν τα χρήματά τους εκεί, να κερδίσουμε αυτή τη μάχη που είναι στοιχείο κλειδί για να έχουμε κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη στο μέλλον, στον κόσμο μας. Άννα Γκόμες τώρα έχει το λόγο, παρακαλώ. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο σε παγκόσμιο επίπεδο Πρέπει να καταπολεμηθεί το σκάνδαλο αυτό, το σκάνδαλο της διαφθοράς, το σκάνδαλο των ποινικά κολάσιμων δραστηριοτήτων. Είναι απαραίτητο η πολιτική, τα πιστοτικά ιδρύματα, οι σύμβουλοι, οι δικηγόροι να μην κρύβονται και κλέβουν τους πολίτες με τέτοιο τρόπο. Η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύει τις εκθέσεις αναχώρα σε σχέση με τις έπαφες ε, τους με τις πολυεθνικές και όχι μόνο οι ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά διεθνή καταπιστεύματα σε άλλες χώρες προσβάσιμα όμως στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί επίσης και η ε, οδηγία για την ανακύκλωση του βρώμικου χρήματος. και είδαμε τι συνέβη και με την Ολλανδία σε σχέση με τη δική μου χώρα, την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπερές, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι, είστε υπεύθυνο για ένα θέμα στο οποίο δεν έχει υπάρξει πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω με τη δική σας όθηση και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως ξεκινήσαμε να το κάνουμε με την υποστήριξη όλων αυτών που καταγγέλουν των δημοσιογράφων, των απλών πολιτών να κινητοποιηθείτε έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το σκάνδαλο. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι θα σας υποστηρίξουμε και να σας πούμε ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετατρέψει την ειδική της Επιτροπή σε ερευνητική επιτροπή ο στόχος θα είναι να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας ε, στον κοινό αγώνα. Εμείς λοιπόν επί τη βάση των προτάσεων τις οποίες καταθέτεται και στα πλαίσια επίσης του, των κύκλων και των συναντήσεων της ομάδας των 20 θα πρέπει ισότιμα με τους εταίρους μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών σε έναν τομέα στον οποίο τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αφήσαμε τις πολυεθνικές να καθορίζουν το παιχνίδι. Ezzel képviselőtársaimmal a végére értünk Στο τέλος, της, ε, συζήτησης περνάμε στο ΚΕΤΣΙΑ τον λόγο έχει ο κ. Τόμ και ήταν πάρα πολύ αυστηρή στο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως το θέμα αυτό με τα έγγραφα του Παναμά είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι και κάτι καινούριο ταυτόχρονα. Έχουμε λάβει πάρα πολλά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμφωνίες με τρίτες χώρες ε, κτλ. αλλά προφανώς αυτά δεν επαρκούν χάνονται δισεκατομμύρια λεφτά τα οποία θα πηγαίνανε στα σχολεία, στις εργασίες, στα παιδιά μας. Η φοροδιαφυγή και η απόκρυψη του πλούτου είναι απαράδεκτη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πιο σοβαρά αυτήν την υπόθεση. Γιατί είναι τόσο ελκυστική η φορολογική παράδοση, παράδειση. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Ε, γιατί είναι τόσο ε, δυσάρεστα τα δικά μας φορολογικά συστήματα. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καπούτο για ένα λεπτό. Νομίζω ότι μιλάμε για μια μεγάλη ζημιά στη σταθερότητα του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Απαιτείται να υπάρχει μια φυσική διαφάνεια στις συναλλαγές της οικονομικές και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πρωτοπόρο στη διεθνή οικονομική διακυβέρνηση. Πρέπει να δράσουμε το ταχύτερο δυνατόν και στον φορολογικό τομέα και να καταστούμε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Οι εκθέσεις ανά χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να συνοδευτούν και από άλλες διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν την διαφυγή των κερδών προς χώρες με χαμηλότερα φορολογικά συστήματα. Θα πρέπει επίσης να ελεγχθούν καλύτερα οι επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητες σε πολλαπλές χώρες και περιοχές. Μαρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν χρειαζόταν τα Panama Papers για να μάθουμε ότι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που παράγουν υπερκέρδη φοροδιαφεύγουν μέσω των ενδοομιλικών συναλλαγών και άλλων τρίκ και αποκρύπτουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους. Άλλωστε οι ειδικοί υπολογίζουν το ποσό των κεφαλαίων που τοποθετούνται σε αυτά τα κράτη από 7 έως 23 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, είτε από 10 έως 30% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος στην ευρωπαϊκή ένωση οι απώλειες λόγω εταιρικής αποφυγής μέσω μεταφοράς κερδών υπολογίζονται σε 50 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. από τα αρχεία που διέρευσαν στον τύπο φαίνεται ότι στις πρακτικές φοροδιαφυγής συμμετείχαν κυρίως εταιρείες του τραπεζικού τομέα όπως η societe generale και η deutsche bank αλλά και άλλες εταιρείες που έχουν απασχολήσει τη δικαιοσύνη κατά το παρελθόν όπως η siemens για τις δίθεν επενδύσεις των ευρωπαϊκών εταιριών σε τρίτες χώρες υπεύθυνη είναι η ευρωπαϊκή ένωση. ήρθε καιρός να δημιουργηθεί ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα χωρίς γκρίζες ζώνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να σταματήσει το φορολογικό ντάμπινγκ των πολυεθνικών εταιριών σε λουξεμβούργο και ολλανδία και να φορολογούνται τα κέρδη των πολυεθνικών στις χώρες όπου αποκομίζονται. ευχαριστώ prevaranti biti brži od nas? do kada će Ευχαριστώ. ότι... ευχαριστώ. πόσο θα παραμείνει έτσι αυτή η κατάσταση, πόσο είναι δυνατόν να ε, αντιστεκόμαστε στη δημιουργία μιας ε, ευρωπαϊκής ε, αρχής πληροφοριών που θα καταπολεμήσει και τον εξτρεμισμό αλλά και τους κλέφτες. Ε, λέμε πως όλα είναι νόμιμα και είναι ένα θέμα φοροαποφυγής. Ε, είναι αδιάφορο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και το θέμα είναι ακριβώς πώς θα έχουμε περισσότερα λεφτά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Επίτροπε, σας παρακαλώ να κινητοποιηθείτε. Έχετε τη στήριξη μας και περιμένουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. ο Χρυσόφωνος έχει το λόγο. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις μέσω Παναμά για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε μαζική κλίμακα καθιστούν εμφανή την ανάγκη αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία και με όσα ε, μη ευρωπαϊκά κράτη αποδειχθούν πρόθυμα να ακολουθήσουν. η ύπαρξη σε διάφορα μέρη της ιφιλίου των λεγόμενων φορολογικών παραδείσων όπου υποθάλπονται όλες οι μορφές του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος αποτελεί διαρκή πρόκληση όταν μάλιστα τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων κατεδαφίζονται στο όνομα της δημοσιονομικής έκτακτης ανάγκης. πρέπει να καταρτιστεί ένας παγκόσμιος κατάλογος των κρατών τα οποία παρέχουν αθέμητα πλεονεκτήματα στα εξωχώρια προέλευση κεφάλαια και να φορολογηθούν όλα τα εμβάσματα προ τράπεζε των κρατών αυτών. πρέπει ακόμα να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των πληροφοριοδοτών ούτω ώστε να διαλευκανθούν τα οικονομικά εγκλήματα. η ώρα για δράση είναι τώρα. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια για την τέταρτη αναθεώρηση των κατευθυντηριών γραμμών για την νομοποίηση παράνομου χρήματος, έχω υποστηρίξει ένα μητρό που να καταγράφονται όλοι οι φορολογικοί παράδεισοι. Αυτό το μητρό είναι αναγκαίο έτσι ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που είναι απλώς ε, ένα, έχουν μια διεύθυνση γραμματοκιβωτίου και δεν υπάρχουν πραγματικά και να μην εξαρτώμεθα τελικά από διαρροές ή από συμπράξεις δημοσιογράφων οι οποίοι ερευνούν τέτοιες υποθέσεις. Ήλπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει με νέε προτάσει για τέτοιε κατευθυντήριε γραμμέ ώστε να αντιμετωπιστεί η νομοποίηση παράνομου χρήματο. Πρέπει να ξαναδούμε αυτή την υπόθεση του Μητρό, γιατί το βασικό είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε, δεν πρέπει να περιμένουμε από τον κύριο Κάμερον αν θα παραδεχτεί, αλλά να υπάρχουν νέες προτάσεις μέχρι την 1η Ιουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ανακάλυψη των ε, εγγράφων αυτών του Παναμά έχουν σαν αποτέλεσμα πολλές χώρες να αρχίζουν έρευνες. Όλοι γνωρίζουμε ότι η νομοποίηση παράνομου χρήματος και η φοροποφυγή είναι κατά των κανόνων που ισχύουν παγκοσμίω. Είναι αλήθεια βέβαια ότι τα προβλήματα τέτοιων ε, που φαίνονται από αυτά τα έγγραφα είναι σαφές. 50-60 εκατομμύρια το χρόνο από την Ευρώπη και μόνο. Η ειδική, στην Ειδική Επιτροπή έχουμε συναντήσει εκπροσώπους πολυεθνικών και έχουμε εξετάσει τις συστάσεις του ΟΣΑ που μιλούν για περισσότερη διαφάνεια και απλοποίηση των φορολογικών κανόνων. Όμως, παραμένει το απόρριτο πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θέλει να κάνει ένα τολμηρό βήμα προς τα μπρος και να απαιτήσει ειδικέ πληροφορίες όσον αφορά το επαγγελματικό απόρριτο. Είναι ένα βήμα παραπάνω, αλλά ελπίζουμε να γίνουν ακόμα περισσότερο πράγματα, εκστρατείε ώστε η διαφάνεια να κυριαρχήσει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκραπίνη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, η νομοποίηση παράνομου χρήματο, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είναι ένα πρόβλημα που ουσιαστικά ταυτίζεται με τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι χώρε μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Είναι θέμα διαχείρισης. Παρόλα αυτά, η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή, η φορολογική παράδειση ανθίζουν όλο και περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν οι χώρε μέλη να μην τα καταφέρνουν από μόνες τους όμως σίγουρα δυσκολεύονται. Οπότε, τι έχουν κάνει οι χώρες μέλη, τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι έχουν κάνει οι διεθνείς οργανισμοί. Είναι τρομερά όσα αποκαλύπτονται από τους δημοσιογράφους στα έγγραφα αυτά του Παναμά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις και νομοποίηση παράνομου χρήματος και εμείς να μην καταφέρουμε να σταματήσουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λέει ο κύριος Ζάνη, φοβούμε ότι αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερες προκλήσεις από ό,τι φαίνεται στη σημερινή συζήτηση. Αυτοί που διαβάζουν τις εφημερίδες, μπορώ να σας πω ότι κι εγώ, αν διάβαζα τις εφημερίδες, δεν θα μπορούσα να φανταστώ μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση που να μην έχει μια offshore εταιρεία ή τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εσόδων της Ευρώπης περνάει αφορολόγητο. Και γι' αυτό ακριβώς είναι που λέμε ότι ένα 1% του πληθυσμού σήμερα έχει όλο τον πλούτο του κόσμου λίγο πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επίτροπε, οι ερωτήσεις ήταν πολλές και προτάσεις όμως και επικριτική. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας λοιπόν. Σας ακούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για μια εξαιρετική συζήτηση που δείχνει ότι σε όλες τις πλευρές της Ολομέλειας υπάρχει επιθυμία για ένα ισχυρό βίαιο αγώνα εναντίον της φοροδιαφυγής και του ξεπλήματος. Τα Panama Papers υπογραμμίζουν για μια ακόμη φορά την ανάγκη για μια καλύτερα συντονισμένη, περισσότερο ισχυρή ε, και πιο σφαιρική προσπάθεια καταπολέμησης των δραστηριοτήτων αυτών όχι μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης αλλά και πέραν αυτές. Έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα τεράστιου μεγέθους, οπότε και οι απαντήσεις οι πολιτικές που θα δώσουμε θα πρέπει να είναι διεθνείς και νομίζω ότι η Επιτροπή μας είναι αποφασισμένη, έχει την δυνατότητα, υπάρχουμε αρκετοί επίτροποι που ασχολούμεθα με το θέμα και οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Στο άμεσο μέλλον λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει, αναλάβει ε, φιλόδοξες πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται στο λεγόμενο pipeline θα παρουσιάσουμε τις νέες τροπολογίες μας στην οδηγία καταπολέμησης του ξεπλήματος μέχρι τον μήνα Ιούνιο. Και αυτό θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το προληπτικό σχέλος θα βοηθήσει την καταπολέμηση των ανώνυμων συναλλαγών και θα καταστήσει την απάντησή μας στην πρόκληση αυτή πιο διαφθρωμένη. Η συνάδελφος άλλωστε Βεραγιούροβα είναι εδώ στη διάθεσή σας για να σας δώσει όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες. Θα επανέλθουμε επίσης και στο λεγόμενο CCCTB, η άξις. Νομίζω ότι και εδώ θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του ε, κατά του ξεπλήματος στο, στην εσωτερική αγορά. Θα παρουσιάσουμε έναν πίνακα ο οποίος θα επιτρέψει νομίζω να δούμε τα καθεστώτα τα οποία ισχύουν στις διάφορες τρίτες χώρες και αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε την λεγόμενη μαύρη λίστα στην οποία έχω αναφερθεί. Και τελικά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους διεθνείς μας εταίρους, την ομάδα των 20, τον ΩΣΑ, τον ΚΑΦΗ, έτσι ώστε οι υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί ε, να ισχύσουν στο σύνολο της Ιφιλίου. Ξέρω ότι οι ανησυχίες μας αυτές τις σημερίζεται και η Ολλανδική Προεδρία η οποία έχει εμπλακεί στην υπόθεση αυτή και προσπαθεί με κάθε τρόπο, το ξέρω και για τον Κέρον Ντάισελμπλουμ, ε, προσπαθεί να φέρει τα κράτη-μέλη μπροστά στις ευθύνες τους και να αναλάβουν ε, να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Θα γίνουν προσπάθειες λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω αυτά, για αυτά τα οποία μας είπατε, να δώσω όμως δύο απαντήσεις, δύο-τρεις απαντήσεις πιο συγκεκριμένες προς τους ευρωβουλευτές τους οποίους εκτιμώ. Είπατε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδρασε νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί παρά να προτείνει και αυτό το έχουμε κάνει. Το κάναμε και στην πρότασή μας ε, για τα tax rulings, για την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο έχει επιταχύνει τις διαδικασίες και νομίζω ότι και τα Panama Papers ε, θα πρέπει να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Αντί να ασκείτε κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργαστείτε μαζί μας γιατί είμαστε σύμμαχοι για τον κύριο Βούλφ με την γνωστή κομψότητά του παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν ένα σύστημα φορολογικών ε, παραδείσων και κατηγόρησε τους 47.000 υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λέγοντας ότι είναι απατεώνες και ότι εμείς είμαστε τα αφεντικά των απατεώνων. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Εμείς πληρώνουμε φόρους αντίθετα με άλλους η ιδέα ενός επιτρόπου ή ενός διεθνούς υπαλλήλου που δεν πληρώνει φόρους είναι εντελώς λανθασμένη και αυτό ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να εξοικονομούμε και χρήματα από το 2014 μέχρι το 2020 θα υπάρξει εξοικονόμηση ε, κατά 4,3 δις ε, ε, χρημάτων για τις διοικητικές δαπάνες και 1,5 περίπου από αυτά θα προέλθουν από μειώσεις αμοιβών. Και ο φόρος ο οποίος πληρώνεται από τους υπαλλήλους είναι από 8% μέχρι 43%. Ποσοστά επιβολής φόρου δηλαδή υψηλότερα από αυτά τα οποία υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Και πληρώνουν φυσικά και τις κοινωνικές τους συνεισφορές. Λοιπόν, σταματήστε όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν χώρες που δεν πρέπει να πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θυμίζω ότι υπάρχουν δύο βουλευτές του UKIP που έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης για φορολογικές δαπάνες ή για καταχρήσεις δημοσίου χρήματος. Λοιπόν, σας παρακαλώ Πρώτον, αυτά τα οποία λέτε είναι λάθος και είναι και πολύ κακόγουστα γιατί θα πρέπει να κοιτάτε να καθαρίσετε τη δική σας αυλή πρώτα και μετά να ασχοληθείτε με άλλους. Τώρα για τον κύριο Λάμπερτς έχω ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον κύριο Λάμπερτς και γνωρίζει το θέμα πάρα πολύ καλά. Μου έθεσε ερωτήσεις αλλά δεν είναι εδώ για να ακούσει την απάντησή μου δεν είναι πάρα πολύ κομψό. Καλό είναι να μπορέσουμε να, μπορέσουμε να συζητήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο και με πλήγωσε αυτά το οποίο είπε. Είπε ότι η τελευταία συνάντηση που είχαμε κάνει ήταν ευχάριστη και τον είχα κάνει να χαμογελάσει. Αλλά αυτό που είπε δεν μου άρεσαν καθόλου. Είπε ότι η Επιτροπή υπόκειται στα διάφορα λόμπι. Αυτό είναι εντελώς λάθος, είναι πραγματικό λάθος. Ε, προηγουμένως έγινε επίσης μία πρόταση οδηγίας για το CVCR το οποίο ξεπερνά αυτά τα οποία προτείνουν οι διεθνείς οργανώσεις. Όταν βλέπετε τις προτάσεις του ΟΣΑ λέει ότι θα πρέπει να ε, γίνει πιο διαφανής η φορολογική ε, μηχανή των κρατών μελών. Νομίζω ότι και στην, στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία και στο εσωτερικό της Ευρώπης τα στοιχεία είναι διαθέσιμα. Ακόμα και για τις διεθνείς συναλλαγές. Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο, οι πρώτοι επαναλαμβάνω στον κόσμο, οι πιο φιλόδοξοι και οι πιο απαιτητικοί. Καταλαβαίνω ότι οι βουλευτές είναι πολιτικοί και θέλουν να κάνουν πολιτική και είναι απαιτητικοί απέναντί μας είναι ευθύνη τους αυτό. Αλλά παρόλα αυτά σας παρακαλώ όταν προσπαθούμε να κάνουμε ένα συλλογικό βήμα, ένα βήμα προόδου που πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση να το αναγνωρίσετε παρακαλώ, να το πείτε και όχι να ονοματίζετε και να κατηγορείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα, είμαστε σύμμαχοι, οι επίτροποι που είμαστε εδώ παρόντες, το σύνολο ε, των Επιτρόπων με τον Πρόεδρό μας που μας στηρίζει συνεχώς. Θέλουμε να είμαστε ηγέτες στον κόσμο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αυτά τα οποία προτείνουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Λάμπερτς είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό και γι' αυτό ακριβώς ε, υποστηρίζω ότι αυτά τα οποία είπε τα είπε με κακή πίστη. Συνεπώς λοιπόν ας συνεργαστούμε και μαζί του και με την ομάδα των Πρασίνων και με όλες τις πολιτικές ομάδες τις οποίες σέβομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν τους ίδιους στόχους. Βασικός στόχος είναι η διαφάνεια, βασικός στόχος είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ας προχωρήσουμε από κοινού και ας μην περιοριστούμε σε στήρες και αντιπαραγωγικές πολεμικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως όλα τα όργανα δεν είναι τέλεια, κανένα όργανο διεθνές δεν είναι τέλειο. Παρ' όλα αυτά δεν έχει σε καμία περίπτωση λόγους να κοκκινήσει για αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή και είναι υπερήφανη για τις προτάσεις της. Είναι βήματα προόδου τα οποία δεν έχουν γίνει από καμία άλλη χώρα στον κόσμο, από καμία άλλη ομάδα χωρών στον κόσμο. Σας eh, eh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μήπως ο συνάδελφο θα μπορούσε, αν μου επιτρέπετε, να προσθέσει κάποια πράγματα. Ασφαλώ, Παρακαλώ. Η κυρία Γιουροβα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να προσθέσω κι εγώ κάποιο σύντομο σχόλιο για να απαντήσω στις ερωτήσεις όσον αφορά την νομοποίηση του παράνομου χρήματος. Ναι, έχετε δίκιο. Πρέπει να υιοθετήσουμε διάφορα μέτρα έτσι ώστε οι αρχές να έχουν περισσότερες εξουσίες για να αντιμετωπίσουν την ε, παράνομη νομοποίηση παράνομου χρήματος και να μπορούν να έχουν στοιχεία για όλα αυτά. Έχουμε ήδη πετύχει σημαντικά αποτελέσματα όμως όσον αφορά αυτό το θέμα με την οδηγία μας για την νομοποίηση παράνομου χρήματος. Μεταξύ άλλων η οδηγία αυτή προβλέπει κεντρικά μητρώα όπου αναφέρεται η ιδιοκτησία. Και τώρα προχωρούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην ενσωμάτωση της νομοθεσίας αυτής στην εθνική νομοθεσία των χωρών μελών. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Έτσι τα μητρώα αυτά θα μπορούν να λειτουργήσουν από το τέλος του 2016. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την ενσωμάτωση αυτή στην εθνική νομοθεσία και εγώ έχω επαφές με τους ομολόγους μου στις χώρες μέλη προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα. Και έχετε επίση δίκιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί τώρα την οδηγία αυτή, όπως αναφέρθηκε ε, στη συζήτηση που κάναμε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την πρότασή μας θα την έχετε μέχρι την 1η Ιουνίου και στόχος μας είναι να εμποδίσουμε τους τρομοκράτες να χρησιμοποιούν χρήματα με ανώνυμες ε, μεταφορές χρημάτων αλλά και άλλους τρόπους που κάνουν τις συναλλαγές τους. Συχνά τέτοιου είδους συναλλαγές είναι η πρώτη ένδειξη για τρομοκρατική δράση που ετοιμάζεται. Τέλος. Στο πρόγραμμα δράσης μας σκοπεύουμε και να εναρμονίσουμε τις κυρώσεις όσον αφορά την νομοποίηση παράνομου χρήματος. Σας ευχαριστώ κυρία Γιούροβα. Συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε δύο επιτρόπους εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα θα δώσω τον λόγο στην ε, Υπουργό, την κυρία Πλασχέρτ, για να μας πει τι έχει να μας πει από το Συμβουλίο. Να σας πω, εν ολίγης, οι αποκαλύψεις μας δείχνουν πως η δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, κατά του ξεβλήματος χρήματος και της φορολογικής απάτης έχει μεγάλη σημασία. Κοινός μας στόχος είναι να την συνεχίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο και το Συμβούλιο θέλει βεβαίως να γνωρίζει τα γεγονότα όσο και εσείς στο Κοινοβούλιο και η Κομισιόν είμαι σίγουρη. Γι' αυτό ακριβώ θα εξετάσουμε τις πληροφορίες, τα έγγραφα αυτά και την πολιτική μας ε, με στόχο να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Είμαι σίγουρη πως όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και είμαι επίσης σίγουρη ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη μάχη και είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε γρήγορα και αποτελεσματικά και καλό όλα τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει στα μέτρα που ε, υπάρχουν επιτάπητος και τα μέτρα τα οποία προφανώς ε, και πιθανότατα θα έρθουν προσεχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Υπουργέ για αυτές τις ε, παρατηρήσεις σας. Έτσι τελειώνει η συζήτηση.